Καλό απόγευμα σε όλους. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Διαμαντούρο, ο οποίος ε, περιβρίσκεται εδώ για την παρουσίαση της ετήσιας εκθεσής του, που θα δούμε αμέσως ε, αφού ολοκληρώσουμε το σημείο 15, δηλαδή τις ανακοινώσεις σχετικά με τις αποφάσεις της συνεδρίασης των συντονιστών. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των συντονιστών αποφασίστηκε σε ό,τι αφορά το διορισμό εισηγητή για την ειδική έκθεση για την κακοδίκηση για το θέμα της επέκτασης του αεροδρομίου της Βιέννης αποφασίστηκε να ανατεθεί στους πρασίνους και κατόπιν σύντομα θα ανακοινωθεί και το όνομα του συναδέλφου της συναδέλφου που θα αναλάβει την εκθέση αυτή. Σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία των πολιτών, στην ομάδα των συντονιστών ε, ξεκινήσαμε τις ε, προετοιμασίες για να περάσουμε στο στάδιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων ε, που ανέλαβε η Επιτροπή μας η ομάδα των συντονιστών αποφάσισε και μέσω της σύγκλησης εκτάκτων συνεδριάσεων των συντονιστών να προβεί σε ένα προβληματισμό που κατόπιν θα παρουσιάσει στους ε, οργανισμούς που θα πρέπει να λάβουν τις συγκεκριμένες αποφάσεις. Ουσιαστικά Ασχοληθήκαμε μεταξύ τα σημεία. Καταρχήν, για να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα ε, για τις έκτακτες συνεδριάσεις, τουλάχιστον τέσσερις έκτακτες συνεδριάσεις ε, μέσα σε ένα χρόνο, για να μπορούν να λάβουν χώρα δημόσιες ακροάσεις που έχουν ανατεθεί και στη δική μας Επιτροπή. Είναι αρμοδιότητα της δικής μας Επιτροπής. Το δεύτερο σημείο είναι να βελτιωθούν τα συστήματα ενημέρωσης μέσω πυλών που σε μεγάλο βαθμό μπορούν να ικανοποιήσουν ε, τις, ε, τα αιτήματα των πολιτών όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Και επίσης σταθήκαμε στην ε, ευκαιρία να διαφοροποιήσουμε μεταξύ των αναφορών και των πρωτοβουλειών των πολιτών, δυνάμει του άρθρου 203α. προβλέπεται αρμοδιότητα της Επιτροπής Αναφορών μόνο εκεί που οι όσοι παρουσιάζουν την πρωτοβουλία των πολιτών αν απορριφθεί αυτή από την Κομισιόν, ζητήσουν οι άνθρωποι αυτοί να υπάρχει μετατροπή της σε αναφορά. Δεν μπορεί η Επιτροπή Δυνάμει Δικής της Πρωτοβουλίας ε, να προβεί σε κάτι τέτοιο. Καθώς πρόκειται για τελώς διαφορετικά έγγραφα. Επίσης, σκεφτήκαμε να κάνουμε μια συζήτηση με όλους όσους εμπλέκονται στην ε, διαδικασία της ανάληψης πρωτοβουλίας πολιτών. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να συναντήσουμε τον κύριο Παπαστάμκο, ο οποίος είναι αρμόδιος και παρακολουθεί τη διαδικασία της πρωτοβουλίας των πολιτών, τον αντιπρόεδρο Σεύκοβιτς και τον πρόεδρο της διάσκεψης των επιτροπών, τον Πρόεδρο των επιτροπών, που είναι ο συνάδελφος ο κύριος Λένε. Έτσι λοιπόν θα σας διατηρούμε ενημερωμένου ε, για τις μελλοντικέ εξελίξεις των δραστηριοτήτων αυτών. Η ομάδα των συντονιστών επίσης αποφάσισε σε κατεπίγουσα διαδικασία να συμπεριλάβει την αναφορά για την, ε, το χώρο υγειονομικής ταφής ε, στο Πιάντελόλμο κοντά στη Ρώμη ε, καθώς ε, οι ίδιοι οι υπογράφοντες, οι ίδιοι αναφέροντες ε, ανέφεραν αυτό το θέμα ως κατεπήγον, σημείο 4. Είχαμε πολλές αναφορές που παρουσιάστηκαν σε σχέση με την εξόριξη σχιστολιθικού αερίου. Οι συντονιστές καθόρισαν ως ημερομηνία για την οργάνωση ενός εργαστηρίου για το θέμα, έτσι όπως συμφωνήθηκε στο παρελθόν, την 9η Οκτωβρίου και θα θέλαμε να συμμετέχουν και οι επιτροπές ΕΝΒΙ και ΙΤΡΕ και να ζητήσουμε και μία συνεισφορά από τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος στο θέμα της οργάνωσης, ε, καθώς ε, πρόσφατα ε, παρακολούθησε ένα σεμινάριο για το θέμα αυτό. Και αυτό το θέμα, όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και αφορά πολλούς πολίτες. Η ομάδα των συντονιστών επίσης ανέκρινε το ερωτηματολόγιο που έχει εκπονηθεί από την ομάδα εργασίας ε, για την Ομοθεσία για την παράκτια ζώνη στην Ισπανία, για τις παράκτιες ζώνες στην Ισπανία. Έχουν ε, ταυτοποιηθεί κάποιες συγκεκριμένε ρωτήσεις κατά τη διάρκεια της ε, συνεδρίασης της ομάδας εργασίας και η ομάδα των συντονιστών για την επόμενη συνεδρία εξέτασε μόνο ορισμένα από τα θέματα που θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης. Αλλά η πρόταση της ημερήσιας διάταξης ε, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, το κείμενο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, θα υποβληθεί στους αδέλφους για τελική, τελική έγκριση και φυσικά θα δυναμηθεί και σε εσά. Και για να κλείσω, να σας ενημερώσω για το εξής. Η συνεδρία τη Επιτροπής Περιβάλλοντος τη Επιτροπή των Περιφερειών θα λάβει η χώρα στι 28 Ιουνίου. Πρόκειται για μια συνεδρίαση πολύ σημαντική και πολύ ενδιαφέρουσα για τη δική μας Επιτροπή που ασχολείται πάντοτε όλο ένα και περισσότερο με περιβαλλοντικά ζητήματα γιατί Στη συνεδρίαση εκείνη θα συζητηθεί το θέμα της εφαρμογής της νέας περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύω ότι η συνεισφορά μας σε εκείνη τη συνεδρία θα μπορούσε να είναι χρήσιμη. Δεν υπήρξε κάποια άλλη ανακοίνωση, ούτε άλλα σημεία προς έγκριση. Και ζητώ εδώ την έγκριση από τους συναδέλφους της Επιτροπής. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, επομένως εγκρίνουμε όσο αποφασίστηκαν και στην ομάδα των συντονιστών. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την ολιγόλεπτη καθυστέρηση κ. Διαμαντούρου. εγώ θα σας δώσω τώρα το λόγο, θα δώσω το λόγο στον κύριο Διαμαντούρο για να μας παρουσιάσει την εκθεσή του. Παρακαλώ. Eh, Ο κύριος ε, Μποστινάρου, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λίγα λεπτά το χρόνο σας θα χρησιμοποιήσω μόνο για να παρουσιάσω ένα βιβλίο το οποίο σας περιμένει στην είσοδο. Είναι ένα ιδιαίτερο βιβλίο. Ένα βιβλίο που αναφέρεται σε ένα ε, μεγάλο έργο εξόριξης χρυσού στη χώρα μου και αναφέρεται και στην ε, βιομηχανία εξόριξης χρυσού και στην ε, βιώσιμη ανάπτυξή της. Το βιβλίο αυτό έχει συνεισφορές από πολλούς Ρουμάνους επιστήμονες, σημαντικές ρουμανικές ΜΚΟ, καθώς και τη συνεισφορά μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίοι αγωνίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο Επίσης παρουσιάζει τις απόψεις ε, ανθρώπων που εμποδίστηκαν από το να μιλήσουν στη χώρα μου. Ήταν θύματα μιας πολύ επιθετικής ε, εκστρατείας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τέλος, στο βιβλίο αναφέρονται τα ε, κοινοτικά πρότυπα τα οποία πρέπει να είναι σεβαστά και να εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βιβλίο είναι επίσης μια πηγή αναφοράς για όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν με την βιομηχανία εξόρυξης χρυσού στην Ευρώπη. Και είναι μια πρόσκληση για να ενημερωθούν και μετά να αποφασίσουν για τον τομέα αυτό. Έπειτα το βιβλίο είναι ένας φόρος τιμής στον αγώνα που έγινε από την ρουμανική κοινωνία των πολιτών η οποία κινητοποιήθηκε με εκπληκτικό τρόπο για να αμυνθεί και να υπερασπιστεί κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ο αγώνας μας και η συμβολή μας έχουν ευρωπαϊκή διάσταση και αυτό θέλουμε να το, να το ξεκαθαρίσουμε. Μετά την δημοσίευση του βιβλίου ήμουν προσκεκλημένος για να παρουσιάσω το βιβλίο σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία και αυτό που θα επιθυμούσα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ισχύουν τα ε, αυστηρότερα δυνατά πρότυπα και να μην είναι η εξαίρεση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για αυτή την αποτίμηση τιμή στην Επιτροπή και σας ευχαριστούμε και για όσα είπατε, αν και ήταν ε, εκτός προγράμματος. Θα ξαναδώσω τώρα το λόγο στον Ευρωπαϊκό Μισολαβητή, τον κύριο Διαμαντούρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την ευκαιρία να σας απευθυνθώ Σχετικά με το θέμα της αιτήσιας εκθεσής μου για το 2011, η έκθεση περιλαμβάνει κάποια στατιστικά στοιχεία και υλικό που αφορά τις καταγγελίες που έλαβα από τους πολίτες, ε, τις ΜΚΟ, τις εταιρείες και άλλους το 2011. Ήδη έχετε λάβει την πλήρη έκθεση στα αγγλικά και στη γλώσσα σας. Η πλήρης ε, έκθεση θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημε γλώσσες από τον Ιούλιο, όπως συνήθως. Έστελα την έκθεση και στον πρόεδρο Σούλτ στις 22 Μαΐου. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι σας ε, ευχαριστώ για τη συνεχή υποστήριξη του Κοινοβουλίου αλλά και αυτής της Επιτροπής των Ευρωπαϊκό Διαμεσολαβητή και μπορώ να συνδέσω ότι θα συνεργαστώ στενά μαζί σας ε, προκειμένου να παρέχουμε στους πολίτες τα μέγιστα δυνατά ωφέλη από τις ευρωπαϊκές συνθήκες για το σεβασμό των δικαιωμάτων μου και θα δράσω στα πλαίσια της εντολής μου που είναι πολύ συγκεκριμένη. Δηλαδή να ερευνήσω καταγγελίες για κακοδίκηση στα ευρωπαϊκά όργανα και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και φορείς. Το έργο μου λοιπόν είναι συμπληρωματικό σε αυτό αυτές τις επιτροπής, ε, αν και η αντίστοιχη ρόλη μας είναι διαφορετική. Η κακοδίκηση περιλαμβάνει κάθε είδους αθέμητης διοικητικής συμπεριφοράς από ε, καθυστερημένη πληρωμή για διάφορα έργα με μέχρι δημοσίευση ε, πληροφοριών ανακριβών μέχρι μία απάντηση σε μία επιστολή. Οι συστάσεις μου δεν είναι νομικά δεσμευτικέ, όμω ε, με την πειθό προσπαθώ να πετύχω την εξέβρεση φιλικών λύσεων έτσι ώστε και οι καταγγέλλοντες και τα ευρωπαϊκά όργανα να είναι ικανοποιημένοι και οι δύο πλευρές. Έτσι λοιπόν οι υπηρεσίε μου μπορούν να είναι πιο ευέλικτες και ταχύτερες από τις δικαστικές υπηρεσίες και ε, για πάρα πολλούς καταγγέλλοντες ε, κάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι εντελώς δωρεάν κατόπιν της παρέμβασής μου τα όργανα και οι φορείς ε, πολύ συχνά ε, έχουν απελευθερώσει έγγραφα, έχουν διορθώσει τις αντικίες και έχουν θέσει τέλος ε, στις διακρίσεις. Σημαντικά θέματα αρχής όπως οι πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων επιλύονται στο πλαίσιο αυτό. Να στραφώ τώρα στις κύριες στατιστικές ε, της έκθεσης. Το 2011 έλαβα 2.510 καταγγελίες ε, από ΜΚΟ, ενώσεις, ε, πολίτες και εταιρείε. Και για να στραφώ στην γεωγραφική προέλευση μπορώ να σας πω Ισπανία και η Γερμανία ε, ήταν η πηγή του μεγαλύτερου αριθμού καταγγελιών, ακολουθούσαν η Πολωνία και το Βέλγιο, αλλά σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού τους οι περισσότερες καταγγελίες προήρθαν από μικρά κράτη-μέλη όπως το Λουξεμβούργο, η Κύπρος, η Μάλτα και η Σλοβενία. Οι βουλευτές θα βρουν λεπτομέρειες για τις καταγγελίες αναχώρα στην ετήσια έκθεση και στα αριθμητικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην επισκόπηση. Εγώ προσπαθώ να βοηθήσω όποιον στρέφεται στο διαμεσολαβητή, ακόμη και στην περίπτωση που καταγγέλων ε, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά μου. Τον Ιανουάριο του 2009 ξεκίνησα έναν οδηγό επίδραση ε, στην σελίδα μου που είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημε γλώσσες και προσπαθεί να βοηθήσει τους πολίτες για να απευθυνθούν στο πιο κατάλληλο φορέα να του βοηθήσει ε, αναφέρεται και στι υπηρεσίε του Εθνικού Διαμεσολαβητή, στα κράτη-μέλη ή σε διάφορου μηχανισμού επίλυση διαφορών που έχουν δεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως ε, είναι ε, το Solvit, το δίκτυο Solvit για τα διασυνοριακά προβλήματα ή το Ευρωπαϊκό Πόρταλ, η Ευρωπαϊκή Πύλη. Ε, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι πολίτες από την αρχή να απευθύνονται στο αρμόδιο όργανο προκειμένου να αποφύγουμε τις καθυστερήσεις ε, και τις αποτεύσεις ε, που αντιμετωπίζουν προκειμένου να βρουν το σωστό θεσμό από μόνοι τους. Ο αριθμός των καταγγελιών ε, που που απευθύνθηκα σε μένα συνέχισε να πέφτει το 2011 κατά 211. Ε, θεώρησα ότι αυτό ε, οφειλόταν στο ότι για πρώτη φορά οι πολίτες χρησιμοποιώντας τον οδηγό μπορούσαν να βρουν την κατάλληλη διεύθυνση. Το 2011 πάνω από 18.000 άνθρωποι έλαβαν συμβουλή μέσω του οδηγού αυτού. Τώρα αν ε, δούμε ε, τον ε, αριθμό των ετοιμάτων μπορούμε να πούμε ότι πάνω από 22.000 πολίτες δέχτηκαν άμεση βοήθεια από τη Διαμεσολαβητή το 2011 επιπλέον. Η στοσελίδα Διαμεσολαβητή έλαβε πάνω από 200.000 ε, επισκέψεις ο αριθμός ε, των ερευνών που ξεκίνησαν το 2011, δηλαδή 396, μας έδειξε μεγάλη αύξηση εκείνο το έτος, ε, δηλαδή 18%. Η τάση αυτή επιβεβαιώνει ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται στον Ευρωπαίδιο Μεσολαβητή και το κάνουν αυτό για τους ορθούς λόγους. Η μεγάλη αύξηση στις έρευνες ε, που ξεκίνησαν είχε ε, οφειλόταν και στι δικέ μου πρωτοβουλίε προκειμένου να γίνουν πιο φιλικέ προ το χρήση. Ε, Φέτο έχουμε μια διαδικασία που επιτρέπει στου καταγγέλλοντε να αποσαφηνίσουν την καταγγελία του στην περίπτωση που δεν έχω πιστεί ότι πρέπει να προσφύγουμε ε, στο να απευθυνθούμε ε, σε ευρωπαϊκά όργανα. 318 καταγγελίες έκλεισαν ε, το 2011 και αρκετές από αυτές κατέληξαν ε, σε θετική επίλυση. Συμφωνήθηκε μια φιλική λύση, δέχτηκε το όργανο μία σύσταση. Δεν βρήκαμε κακοδίκηση σε 64 περιπτώσεις, ενώ βρήκαμε κακοδίκηση σε 74 περιπτώσεις το οργανό δέχτηκε ένα σχέδιο σύσταση, είτε εν μέρη είτε πλήρως σε 13 περιπτώσεις ενώ 35 περιπτώσεις έκλεισαν με ζωτικέ παρατηρήσεις. Σε 39 υποθέσεις έκανα περαιτέρω παρατηρήσεις για να συμβάλλω στην βελτίωση της επίδοση. μια ε, περαιτέρω μείωση των ζωτικών ε, παρατηρήσεων είναι δυνατό επίση επίσης, όμως τα όργανα πρέπει να λαμβάνουν ένα πιο προδραστικό ρόλο στο να επιλύουν τις καταγγελίες και να έχουμε λύσεις από, από που όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Αυτό ωφελεί και τα δύο μέρη. Κατά τα τρία τελευταία έτη οι ζωτικές παρατηρήσεις ε, ήταν πάνω από 34 κατά μέσο όρο, ενώ ο μέσος όρος ε, ήταν 46 στην περίοδο 2006-2008. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, φέτος στην ετήσια έκθεση και πάλι συμπεριέλαβα την έννοια των υποθέσεων των πολύ σημαντικών star cases προκειμένου να δώσω κάποια παραδείγματα παραδειγματικών πρακτικών διοικητικών και προκειμένου να τονίσω ότι ε, τα όργανα πρέπει να λειτουργούν έτσι ώστε να προωθούν και να, βελτι... να προωθούν να χρησιμοποιούν τις βέλτιστες πρακτικές. Τέτοιες 10 ε, υποθέσεις τονίζονται στην ετήσια έκθεση και παρουσιάζεται στο τμήμα 1-5 της έκθεσης αυτής. Η βούληση των θεσμών για να συνεργαστούν με τη διαμεσολαβητή για να έχουμε ομαλή επίλυση ε, αποτελεί μια σημαντική δέσμευση. Επίσης σημειώνω ότι σε κάποιες περιπτώσεις η επικοδομητική στάση των ίδιων των καταγγελόντων ήταν ζωτική σημασίας για να έχουμε αποτέλεσμα ικανοποιητικό για όλους. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο για τα δικαιώματα των πολιτών και για την επίδοση τη δίκη της Ευρωπαϊκής Ένωση, μια μελέτη που ζητήθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διαμεσολαβητή και δημοσιεύτηκε το 2011, ε, το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνηση και εγκατάσταση ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται το πιο σημαντικό δικαίωμα των πολιτών, σύμφωνα με το 48% όσων απάντησαν. Το δεύτερο πιο σημαντικό δικαίωμα είναι το δικαίωμα στην καλή διοίκηση, 33% και ακολουθεί το δικαίωμα ε, καταγγελίας του Μεσολαβητή, 32%. Από την άλλη, 42% όσων απάντησαν είπαν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι με τη διαφάνεια στη δίκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 52% είπαν ότι ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι πολίτες ξέρουν τα δικαιώματά τους και πώς να τα χρησιμοποιούν. Το να καταστήσουμε προτεραιότητα το στόχο πολιτικής ενημέρωσης των πολιτών το Μάρτιο του 2011 ε, φιλοξένησα τη μεγαλύτερη εκδήλωση που διοργανώθηκε από τη για τους stakeholders, όπως προβλέπει και η συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, σημαντικοί ομιλητέ ήταν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κύριος Βαν ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυρία Ντεϊάννα Βαλαβάλε και αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Βιβιάν Ρέντινγκ. Επίσης, το 2011 δημοσίευσε ένα φυλάδιο με τίτλο «Προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος μπορεί να σας βοηθήσει». Αυτή η νέα δημοσίευση προτιλέπει πληροφορίες για μια σειρά μηχανισμών επίλυσης προβλημάτων που είναι διαθέσιμοι σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι υπήρξε μεγάλη ζήτηση για αυτό το φυλάδιο, πολύ μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο φυλάδιο στην ιστορία του θεσμού του διαμεσολαβητή το επίπεδο τη δυσαρέσκεια με τη ίδια διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρησιμοποίησα την ευκαιρία που μου δόθηκε από τον εορτασμό ε, τη. Ε, των διεθνών δικαιωμάτων για να καλέσω την Ευρωπαϊκή Διοίκηση να είναι πιο προδραστική σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια. Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνω έκκληση στου ευρωπαϊκού θεσμού να εθετήσουν ε, χρήσιμα μητρώα επιγραμμικά για τα έγγραφα και σε ό,τι αφορά τις δικές μου υπηρεσίες στις αρχές του 2011 άρχισα να δημοσιεύω στην ιστοσελίδα μου πληροφορίες για νέες έρευνες μόλις ξεκινούσαν. Αυτή είναι πρακτική διευκολύνει τους πολίτες να παρατηρήσουν πώς προδεύουν από την αρχή πώς προδεύουν οι έρευνες αυτές. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, το 2009 Υιοθέτησα μία δήλωση αποστολή για το θεσμό του Μεσολαβητή που λέει το εξή. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητή ε, σε σχέση με τα ε, θαρρύνει τη διαφάνεια και προωθεί την διοικητικό πολιτισμό των υπηρεσιών, ε, θέλει να οικοδομήσει εμπιστοσύνη μέσω του διαλόγου των πολιτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να προωθήσει ψηλά πρότυπα συμπεριφορά στου θεσμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να έχουμε καλύτερη εφαρμογή της δήλωσης αυτής. Το 2010 υιοθέτησα μια στρατηγική που αποτελεί τη βάση για τις πρωτοβουλίες μου και τις δραστηριότητές μου κατά τη σημερινή μου εντολή. Τα κύρια σημεία στρατηγική αυτή περιλαμβάνουν καταρχήν ενδυνάμωση του συνεχιζόμενου διάλογου με του καταγγέλλοντε στην κοινωνία των πολιτών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, σύμφωνα με τι κεντρικέ δεσμεύσει που αναγράφονται στη συνθήκη τη Λισαβόνα. Δεύτερον, να εντοπίσουμε τι βέλτιστες πρακτικές ε, στο ευρωπαϊκό δίκτυο του διαμεσολαβητή και τρίτο να προωθηθεί ο ρόλος του διαμεσολαβητή στο να προωθηθεί μια διοικητική, ένας διοικητικός πολιτισμός των υπηρεσιών ε, στα ευρωπαϊκά όργανα προκειμένου να έχουμε καλή δίκηση συνεχώς ένα κύριο στοιχείο ε, του να είναι και φιλικό προς τους πολίτες ε, τα όργανα και οι θεσμοί θα πρέπει να προωθήσουν ένα πολιτισμό παροχής υπηρεσιών στους πολίτες προκειμένου να υπάρξει ένα τέτοιο πολιτισμό, ενθαρρύνεται τα μέλη του προσωπικού όχι μόνο να σέβονται την καλή διοίκηση ω νομικό δικαίωμα, αλλά να είναι και ευγενικοί και να συνεργάζονται με του πολίτε, να, θέλουν να ε, εξηγήσουν τι δραστηριότητέ του και το σκεπτικό του και να είναι έτοιμοι να δεκτούν δημόσιο έλεγχο τη συμπεριφορά του. Με τις σκέψεις αυτές κατά νου κατέληξα στο συμπέρασμα ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει μια σύντομη δήλωση σχετικά με αυτέ ε, τι αρχέ που θα μπορούσε να βελτιώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στι ευρωπαϊκέ υπηρεσίε και στου ευρωπαϊκού θεσμού. Σα ενημέρωσα για την πρόθεσή μου προ αυτήν την κατεύθυνση πέρσι και προχώρησα στην κατάρτιση μια τέτοια δήλωση ε, ε, που θα έπρεπε να αντικατοπτρίζεται η συμπεριφορά ε, των δημοσίων υπαλλήλων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκειμένου αυτό να ληφθεί υπόψη στα κράτη-μέλη, ζήτησα ε, κάποιε απόψει από του συναδέλφου ε, στα κράτη-μέλη. Και όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία, ξεκίνησα μια δημόσια διαβούλευση για τις αρχές αυτές το Φεβρουάριο του 2011. Η δημόσια διαβούλευση έμεινε ανοιχτή μέχρι τον Ιούνιο για συνεισφορές και έλαβε 56 πολύτιμες συνεισφορές. Δημοσίευσε μια έκθεση για τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων τον Νοέμβριο που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μου. Σήμερα, σήμερα το πρωί δημοσίευσα τις αρχές ε, της δημόσιας δίκης, θα τις αναφέρω. Πρώτη αρχή. Δέσμευση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες. Οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν πλήρη συνείδηση ότι τα όργανα υπάρχουν για να εξυπηρετούν την Ένωση και τους πολίτες και για να πληρούν τους στόχους της συνθήκης. Πρέπει να κάνουν ε, συστάσεις για να εξυπηρετούν μόνο αυτά τα συμφέροντα πρέπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Και αυτό έχει να κάνει με την δημόσια εμπιστοσύνη και δίνει το παράδειγμα σε άλλους. Δεύτερη αρχή, ακεραιότητα. Οι δημόσιοι πάλι πρέπει ε, να ε, έχουν ευπρέπεια και να συμπεριφέρονται με τρόπο που να επιδέχεται δημόσιο έλεγχο. Αυτή η υποχρέωση δεν εκπληρώνεται μόνο δρώντας σύμφωνα με τον νόμο. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θα πρέπει να έχουν οικονομική υποχρέωση που θα μπορούσε να τους επηρεάσει στην διεκπαιρέωση της υπηρεσίας τους ε, και δεν θα πρέπει να λαμβάνουν δώρα. Δεν θα πρέπει να έχουν ιδιωτικά συμφέροντα αντίθετα με την λειτουργία τους. Θα πρέπει να αποφεύγουν την σύγκρουση συμφερόντων και την εμφάνιση, την παρουσίαση τέτοιων σύγκρουσεων ε, και η υποχρέωση που έχουν ε, ισχύει ακόμα και μετά το τέλος της θητείας τους. Θητείας τους. Τρίτη αρχή, αντικειμενικότητα. Πρέπει να είναι αντικειμενικοί, ανοιχτόμυαλοι, να αναζητούν αποδείξεις και να ακούν διαφορετικές γνώμες, να διορθώνουν ε, τα σφάλματα εκεί όπου υπάρχει συγκριτική αξιολόγηση θα πρέπει να βασίζουν τις αποφάσεις και τις συστάσεις όχι μόνο ε, στα χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τον νόμο αλλά μόνο στην αξία τους, ε, στα, στα πλεονεκτήματα. Δεν θα πρέπει να βασίζονται σε συμπάθεια και αντιπάθεια προς ένα άτομο τέταρτη αρχή σεβασμός των άλλων. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να σέβονται τους άλλους και τους πολίτες, να είναι ευγενικοί, να είναι συνεργάσιμοι και πρόθυμοι, να καταβάλουν πραγματικές προσπάθειες για να κατανοούν τι λένε οι άλλοι και να εκφράζονται σαφώς, με γλώσσα σαφή και ευκρινή. Πέμπτη αρχή διαφάνεια θα πρέπει να εξηγούν τις δραστηριότητές τους και να δίνουν τα αίτια των ε, δραστηριοτήτων τους και να συμμορφώνονται με όλες τις αρχές των δημοσίων υπαλλήλων. Ε, κυρία Πρόεδρε, αξιότυπα μέλη, όπως επανειλημμένα έχω πει, αυτές οι αρχές δεν είναι ούτε ε, η πρώτη ούτε η τελευταία λέξη για τα δεοντολογικά πρότυπα που ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους. Όπως μας έδειξαν οι δημόσιες διαβουλεύσεις, οι κανονισμοί και η καλή ε, συμπεριφορά του διαμεσολαβητή περιλαμβάνουν ε, ρητός και ε, με τρόπο υπονοητό αυτές τις αρχές. Στόχος δεν ήταν να αναπτύξουμε νέα ηθικά πρότυπα, αλλά να αναδείξουμε ε, τι, τι περιμένουν από τους δημοσίους υπαλλήλους και τι περιμένουν οι πολίτες. Προσπαθούμε να είναι όλα ρητά, ούτω ώστε να υπάρχει επικοδομητική συζήτηση ανάμεσα στους δημόσιους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους και ε, το κοινό για το ποια δεοντολογία είναι η κατάλληλη οι διαβουλεύσεις κατέδειξαν την αξία μιας τέτοιας συζήτησης. Δεν προσπαθούμε να επαναλάβουμε αρχές, να συμπληρώσουμε, να υποκαταστήσουμε αρχές, αλλά θέλω να είμαι μια πλούσια πηγή ιδεών από την οποία θα αντλήσω στην συνεργασία μου με τα όργανα στο μέλλον ούτως ώστε να αναπτύξουμε την θεσμική κουλτούρα που θα επιτρέψει την υλοποίηση αυτών των αρχών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Διαμαντούρο για την ε, έκθεσή του και σας ευχαριστούμε για τη δραστηριότητα που καθημερινά στην υπηρεσία που συντονίζετε δεν είναι εύκολο το καθήκον σας και εμείς ε, ως ε, τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου που προστατεύει την ε, δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος της ηθαγένειας από την πλευρά των πολιτών γνωρίζουμε πόσο βαρύ είναι το καθήκον αυτό. Και Βεβαίως, ε, στα πλαίσια της ε, επόμενης συζήτηση για την έκθεση που θα παρουσιάσω ε, και εγώ, θα αναφερθούμε και στη δική σας έκθεση. <clears throat> Στη συνεδρία της 12 Ιουλίου. Ήδη έχουμε στη διάθεσή μας κάποιες ιδέες, μπορούμε να βασιστούμε και στη μεθοδολογική εμπειρία του Ευρωπαϊκού Διαμεσολαβητή για να βελτιώσουμε τη διάρθρωση της δικής μας οργάνωσης και την εκπόνηση των εργασιών μας. Τώρα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νίμαν Κρίστενσελ. Παρακαλώ. Uh, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Διαμαντούρο, τον διαμεσολαβητή μας. Ε, όπως ε, ήθιστε, η Κομισιόν θα ήθελε να απαντήσει. Βρίσκομαι εδώ εκπροσωπεύοντας το όργανο που είναι αρμόδιο για τα περισσότερα... για τα περισσότερα θέματα. Το έργο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή δεν είναι να λαμβάνει νομικά δεσμευτικές αποφάσεις, αλλά να εμπνέει και να, να ηγείται προς μια καλύτερη δημόσια διοίκηση. Είναι μια ηθική αρχή και θα ήθελα να αρχίσω λέγοντα εκ μέρου της Ευρωπαϊκή Επιτροπής ότι η έκθεσή σας πραγματικά ε, δείχνει πόσο εξαιρετική δουλειά έγινε για την επίτευξη του στόχου αυτού και πραγματικά μας ε, οθεί να κάνουμε καλύτερη δουλειά μέρα με τη μέρα. Ε, χαίρομαι πολύ για τα επόμενα χρόνια συνεργασίας μας και φυσικά δεν θα υπάρξει τέλος σε αυτό το έργο. Αυτό το έργο συνεχίζεται και ζούμε σε μια εποχή όπου οι πολίτες και τα θεσμικά όργανα συνδέονται, διαδρούν και η προσπάθεια για να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες ε, θα είναι άιναη. Και Φυσικά νομίζω πως ε, μιλώ και εκ μέρους όλων των άλλων θεσμικών οργάνων και όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν λέω ότι θα χρειαστούμε την συνδρομή σας και στη συνέχεια. Εμείς πιστεύουμε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας που είναι σχετικά πρόσφατη ακόμα και η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, ε, ήταν ένα σημαντικό βήμα στην θέσπιση του, κάθε, του ότι κάθε ίδρυμα πρέπει να διασφαλίζει την σωστή διοίκηση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και πραγματικά καλωσορίζουμε την προσπάθειά σας να δώσετε σάρκα και ώστα σε, αυτά τα, σε αυτούς τους ε, αφηρημένους όρους. Η σχέση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ επικοδομητική και πραγματικά ε, μας ε, χαροποιεί το γεγονός ότι ε, η σχέση αυτή εμβαθύνθηκε τα τελευταία χρόνια. Πραγματικά χαιρόμαστε πολύ για την συνέχιση της συνεργασίας μας τα επόμενα χρόνια. Θα ήθελα να αναφέρω ενώπιόν σα ότι έγιναν εξαιρετικά καρποφόρες ανταλλαγέ τον Φεβρουάριο ανάμεσα στο Σώμα των Επιτρόπων και στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή αλλά και ανάμεσα στους ε, γενικούς διευθυντές. Δεν ήταν τυπικό, τυπική διαδικασία, ήταν πραγματικά μία συζήτηση όπου οι συνάδελφοί μου ανέπτυξαν τις ανησυχίες τους και έτσι διεξήχθη ένας ουσιαστικός διάλογος για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ε, απόδοσή μας, πώς μπορούμε να δουλέψουμε καλύτερα. Φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει το όργανο το οποίο ε, είναι αρμόδιο και έχει άμεση επίπτωση στους πολίτες. Και οι αναφορές στον Ευρωπαϊκό Διαμεσολαβητή υπάγονται στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και να πω ότι το 50% των ε, αναφορών το 58% μάλιστα των αναφορών αυτών. Είναι κάπως, ένα ποσοστό κάπως χαμηλότερο από την περασμένη χρονιά δεν μπορώ να σας πω ότι, κάνουμε, ότι έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, όμως γενικά όσον αφορά τον όγκο εργασία, πιστεύουμε ότι αυτό το 58% είναι ένα ρεαλιστικό ποσοστό και ε, μπορεί να και αντικατοπτρίζει τις ε, αποφάσεις που λαμβάνουμε για τους πολίτες μας. Η Κομισιόν παραμένει δεσμευμένη να ε, εργάζεται με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα για το καλό των πολιτών και να έχει μια διοίκηση καθόλου ανεξάρτητη. Συνεχίζουμε να προσπαθούμε να ενημερώνουμε τους ε, αξιωματούχους μας για τις, ε, για, σχετικά με θέματα δεοντολογίας. Και θα φροντίσω να συνεχίζουν, να συνεχίζε, να ενημερώνονται. Διότι πραγματικά προσπαθούμε για μια αντικειμενική δημόσια διοίκηση και προσπαθούμε να, να ε, κάνουμε την γραφειοκρατία πιο κατανοητή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναλύουμε τα πράγματα, να μην λέμε ότι αυτό είναι ή δεν είναι ηθικό. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς αυτό εφαρμόζεται στην πράξη, πώς, ε, τι σχέση έχει με τον έξω κόσμο. Και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπενθυμίζουμε στους πολίτες τα δικαιώματά τους. Πραγματικά λοιπόν καλωσορίζουμε τον κατάλογο των ε, αρχών υπηρεσιών σε έναν το πολυ, πολυπολιτισμικό κόσμο. Η κυρία Άουκιν, για παράδειγμα, έχει μια διαφορετική ε, αντίληψη από συναδέλφους από άλλα κράτη-μέλη. Ο καθένας το αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Είναι γι' αυτό λοιπόν πάρα πολύ καλό να μας, να μας υπενθυμίζετε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό ξανά θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω, κυρία Διαματούρο, για την ε, πραγματικά εξαιρετική προσπάθεια και θα ήθελα να πω ότι η έκθεσή σας αυτή δείχνει ότι εάν δεν υπήρχε ο θεσμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή θα έπρεπε να τον εφεύρουμε. Διότι πρέπει να υπάρχει κάποιο να μα θυμίζει τα καθήκοντά μα, γιατί κάθε μέρα είμαστε τόσο απασχολημένοι με τη γραφειοκρατία που χρειαζόμαστε κάποιον να μας, να μας υπενθυμίζει τη δουλειά μας, το καθήκον μας. Και αυτό είναι αυτό που εσείς και το επιτελείο σας κάνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Grazie. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας και κυρίως για το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξατε και για την γραμμή που δεν ήταν τόσο αμυντική αλλά παροτριντική που δώσατε. Και ουσιαστικά η Κομισιόν έχει καθήκον να μέσω το δυνατόν καλύτερο τρόπο στις καταγγελίες των πολιτών ε, και σας ευχαριστώ που αναφερθήκατε στο ότι επιθυμείτε τη βελτίωση των επιδόσεων και ελπίζω οι επιδόσεις ε, να βελτιωθούν και κατόπιν των δικών μας συστάσεων της δικής μας Επιτροπής. Συνάδελφος Σονκλέρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω τρεις ερωτήσεις. Καταρχάς, μία τεχνικής φύσεως για τα νούμερα. Ε, εδώ θα ήθελα να, να σας ρωτήσω τι σημαίνει το other, το άλλα και τι σημαίνει το not known. Θα ήθελα να ρωτήσω, να μας δώσετε κάποια παραδείγματα για το τι σημαίνουν αυτά τα σημεία. Έπειτα, για την πληροφόρηση των πολιτών για το έργο σας, για τις ε, για τη δυνατότητα που έχετε να εξετάζετε ένα ζήτημα. Πώς μπορείτε να μεταδώσετε την πληροφορία αυτή στους πολίτες. Ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, βρισκόμαστε πολύ χαμηλά στη λίστα των ε, αναφορών. Και το επίπεδο δυσαρέσκειας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα είναι εξαιρετικά υψηλό πολύ πιο υψηλό από αυτό που φαίνεται σε, αυτό, σε αυτά εδώ το, τα στατιστικά στοιχεία. Πώς σκέφτεστε να αυξήσετε την ενημέρωση των πολιτών. Έχετε σκεφτεί πώς να χρησιμοποιήσετε τους ευρωβουλευτές, να τους καταρτήσετε και ίσως αυτό τους βοηθήσει να δουλέψουν επιτέλους και λίγο. Επίσης πραγματικά με χαρά άκουσα ότι ε, θα υπάρξει περισσότερη διευκρίνηση, αλλά έχω μια ερώτηση σχετικά με την Επιτροπή Προπολογισμού. Διότι σύμφωνα με την έκθεση αυτή, μα λέτε ότι από τα 2.510 αναφορέ το 2011, μόνο 698 υπέπεπταν στι αρμοδιότητέ σα. Όμω εδώ η έκθεση λέει ότι αυξήθηκε ο προπολογισμό σα, που νομίζω ήταν λίγο κάτω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Εάν δούμε πόσες από αυτές τις αναφορές ήταν αρμοδιότητά σας, τότε βλέπουμε ότι υπήρχε μία αύξηση 3,89%. Επίσης, πρόσεξα ότι θέλετε να αυξήσετε τις, τις 8 υφιστάμενες θέσεις. Και πραγματικά θα ήθελα να ακούσω την απάντησή σας. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το όργανο που κηρύσσει την λιτότητα, αλλά δεν το βλέπουμε αυτό στον προπολογισμό. Ευχαριστώ. Κύριε Όκελ. Yes, uh, thank you very much. Ευχαριστώ, πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. για την εισαγωγή σας. Ε, γενικά, όταν βλέπω τον ε, κατάλογο των ε, προσφυγών, τα ποσοστά, Πολλές φορές το λέμε εδώ σε μια επιτροπή, όταν έχετε πολλές προσφυγές από μια χώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι η κατάσταση σε αυτή τη χώρα είναι πάρα πολύ κακή. Θα μπορούσε να είναι καλή η κατάσταση και όπου οι πολίτες είναι ξύπνοι ε, και ενδιαφέρονται Βλέπουμε την Ρουμανία, την Βουλγαρία, είναι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις και νομίζω ότι αυτό ισχύει και γι' αυτό που βλέπουμε εδώ σε αυτή την Επιτροπή, ότι δηλαδή έχετε μια κοινωνία πολιτών πολύ συνειδητή σε ορισμένες χώρες, ενώ η κατάσταση στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία είναι διαφορετική και θα μπορούσα να πω ότι έχουμε πολλές προσφυγές, βλέπουμε, από την Ελλάδα ε, δεν θέλουμε. Αλλά πού είναι, πού είναι όταν ξέρουμε τι συμβαίνει για πάρα πολλά πράγματα. Ε, καμιά φορά λέω στους Ισπανούς συναδέλφους ότι δεν πρέπει να είναι τόσο οργισμένοι που η Ισπανία είναι τόσο συχνά στην ημερήσια διάταξη εδώ. Ε, αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες συμμετέχουν και βλέπουμε τι γίνεται δεν, ε, γενικά αυτό για τον αριθμό των προσφυγών σε μια χώρα. Αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε όλοι και ε, να, να δούμε γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Δεύτερον, σχετικά με τις αρχές ως προς τις δημόσιες υπηρεσίες. Σήμερα το πρωί στην Επιτροπή μας πέρασε η γνωμοδότησή μου για τον νόμο των διοικητικών διαδικασιών στην Ευρώπη. Είναι μια γνωμοδότηση και εκεί ορίσαμε ε, αρχές για τις υπηρεσίες και, και ελπίζω να μπορέσουμε να περάσουμε από τον ήπιο νόμο ε, και έχουμε βεβαίως όλα αυτά τα ωραία λόγια, τις ωραίες προθέσεις από την Κομισιό ε, για το πόσο καλοί θα είμαστε διαφανείς κλπ. κλπ. Όταν προσπαθούμε ε, να έχουμε μυστικοπάθεια, να συγκαλύπτουμε. Φανταστείτε ε, να βγούμε από την νομική βάση της συνθήκης της Λισαβόνας. Οι κανονισμοί για το θέμα αυτό τι γίνεται. Ελπίζω ότι σε συνεργασία και είναι καλό να δουλεύουμε με τους Έλληνες κατά των Δανών για να καταστήσουμε ε, τον κανονισμό αυτό ασφαλέστερος, ούτως ώστε ε, να μην έχουμε να ε, ασχολούμεθα με τους κανόνες ήπιου δικαίου που καμιά φορά δεν έχουν να κάνουν με την πραγματικότητα. Και θα πρόσθετα επίσης αυτό που θα πρέπει εσείς να τονίσετε επίσης, ότι είναι μια εμπειρία από τη Δανία, την Σουηδία, κυρίως τη Σουηδία, όπου έχετε τέτοιες αρχές και όπου και η ίδια η δίκηση επωφελείται, όχι μόνο οι πολίτες, αλλά η ίδια η δίκηση, οι αρχές επωφελούνται, βρίσκονται σε, ένα, σε μια κατάσταση ασφαλέστερη όταν διεκπεραιώνεται η εργασία με αυτές τις αξίες. Και θα ήταν πάρα πολύ καλό αν μπορούσαμε να πείσουμε τους συναδέλφους στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο ότι δεν πρέπει να φοβούνται τόσο πολύ ε, να, να φοβούνται τόσο πολύ τους πολίτες, να εστιάζονται στους πολίτες. Δεν πρέπει τόσο να φοβούνται ε, την διαφανή δημοκρατία. Ίσως ε, δημιουργήσει μια καλύτερη κοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτές τις συμμαχίες αν έχουμε έναν καλό ε, διοικητικό νόμο, μια νομοθεσία ως αποτέλεσμα. Θα ήταν καλό ακόμα και αν ε, δεν μπορείτε να βελτιώσετε την πρόσβασή μας ε, σε έγγραφα. Ευχαριστώ κύριο Σαλαβράκος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα επενέσω τον κύριο Διαμαντούρο. Πρώτα γιατί η έκθεσή του είναι πολύ κατατοπιστική και η ανάλυση του έργου του εξαιρετική, όπως ομολόγησε και ο κύριος εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ε, θέλω να πω ότι τον έκρινα με ιδιαίτερη αυστηρότητα γιατί καταγόμεθα από την ίδια χώρα. Και μάλιστα ο κύριος Διαμαντούρης ήταν ε, για μερικές μέρες ένα όνομα που έπαιζε για πρωθυπουργός της χώρας μας. Είναι ένδειξη του καλού Έλληνα και ξέρετε ε, είμαι από εκείνους που πιστεύω ότι όλα τα κράτη έχουν τους καλούς και τους κακούς και είμαι εναντίον όλων των γενικεύσεων που γίνονται αυτή την εποχή ιδιαίτερα σε μερίδα του ευρωπαϊκού τύπου σχετικά με τη γενίκευση χαρακτηρισμών εις βάρος λαών όπως είναι η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία. Πρόσφατα μάλιστα, δράτω με τις ευκαιρίες να το θίξω εδώ, μια εφημερίδα γερμανική, η Bild, είπε ότι οι Έλληνες ώψη των εκλογών μπορούν να ψηφίσουν οποιοδήποτε δεξιό ή αριστερό καραγκιόζι αλλά είναι δικά μας τα λεφτά. Ε, έχουν, καραγκιόζης είναι μια φιγούρα που είναι καταφρονεμένη ενός κακού ανθρώπου τεμπέλη ο οποίος ζει εις βάρος των άλλων. Καραγκιόζηδες δυστυχώς έχουμε σε όλα τα κράτη και ιδιαίτερα στο κράτος το οποίο αυτή η εφημερίδα κυκλοφορεί. Μάλιστα οι καραγκιόζηδες οι Έλληνες είναι καλοσυνάτοι και ποτέ δεν έχουν γεμίσει με αίμα την Ήπειρο. Αυτοί έχουν καραγκιόζιδες που γεμίσανε με αίμα μια Ήπειρο. Αυτό είναι μια παρένθεση την οποία κάνω γιατί αισθάνομαι ότι σαν Έλληνας και σαν Ευρωπαίος ιδιαίτερα πολίτης δεν πρέπει ο ένας να εξτομίζει εναντίον του άλλου τέτοιους χαρακτηρισμούς. Υπάρχουν καλοί Γερμανοί και κακοί Γερμανοί, καλοί Έλληνες και κακοί Έλληνες, καλοί Ισπανοί και κακοί Ισπανοί, αλλά οι γενιγεύσεις πρέπει να λείψουν. Θέλω να πω το εξή. Ε, εξαρμοδιότητος ο Όμπουσμαν, ο Ευρωπαίος Μεσολαβητής, καλείται μαζί με τις άλλες θεσμικές εξουσίες της κοινότητα να αποκαταστήσει το αίσθημα της δικαιοσύνης προς τον πολίτη. Το αίσθημα δικαιοσύνης είναι πολύ ευρύτερο από την απονομή δικαιοσύνης. Διότι η απονομή δικαιοσύνης αφορά συγκεκριμένη περίπτωση. In concreto, όπως λέγανε στην ε, ε, ε, λατινική γλώσσα. Το αίσθημα όμως δικαιοσύνης είναι in abstracto, είναι γενικό. Και πάνω στο αίσθημα δικαιοσύνης δημιουργούνται οι ισορροπίες των λαών. Οι λαοί δέχονται να μειωθεί ο τρόπος ζωής τους δέχονται να υποστούν θυσίε αρκεί να αισθάνονται ότι η κατανομή αυτών των θυσιών γίνεται μέσα σε ένα πλαίσιο δικαιοσύνης. Και σε αυτή την περίοδο που όλη η Ευρώπη και ιδιαίτερα ο Νότος, κύριε Διαμαντούρο, έχει ένα πρόβλημα κοινωνικής αναταραχής λόγω της κρίσης της οικονομικής που υπάρχει, αντιλαμβάνεστε ότι η αποκατάσταση του αισθήματο δικαιοσύνης και από το θεσμό το δικό σας είναι ένα σημαντικό φορτίο και αναμένει ένα σημαντικό έργο. Σας εύχομαι και το ελπίζω το έργο αυτό να το φέρετε σε πέρας. Εκείνο το οποίο έχω να πω σε σχέση με τον προϋπολογισμό τον οποίο είδα διεπίστωσα ότι πράγματι έχετε 3,89 μια αύξηση του προϋπολογισμού και τον ανέλησα ότι προφανώς οφείλεται σε αύξηση των αμοιβών προσωπικού κατά 113.000 ευρώ και των εξόδων μετεγκαταστάσεώς σας διότι ε, το κτίριο στο οποίο στεγάζεστε τώρα απεφασίστη να γίνει μουσείο. Επομένως δεν ευθύνεται από ό,τι αντελήφθη ε, σε δική σας αλόγιστη δαπάνη ή δική σας υπέρβαση της, ε, του προϋπολογισμού και θα ήθελα να το αποκαταστήσω σε αυτή τη φάση. Πιστεύω ότι όλοι μας σε αυτή την αίθουσα με τους θεσμούς στους οποίους στην ουσία δίδεται ε, μια ρομαντική σημασία διότι οι θεσμοί οι οποίοι δεν επιβάλλονται δεν έχουν την δυνατότητα αποφάσεων εκτελεστών η διάσταση είναι ρομαντική και πρέπει να υπάρχει αυτός ο ρομαντισμός για να ισορροπήσουμε όπως είπα τις κοινωνίες διότι κάποιος θα έπρεπε να είναι πάντα πίσω από κάθε άλλον και κάποιος να παρακολουθεί τον άλλον, να τον αστυνομεύει. Και το μεγάλο ερώτημα του Κικέρο να ήταν ποιος θα παρακολουθεί τους παρακολουθούντες. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να συνεχίσετε να πηγαίνετε καλά. Ευχαριστούμε κυρία Μπουλάρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ευρωπαϊκό Μεσολαβητή για το σύνολο του έργου του και για τον επικοδομητικό του ρόλο ω οδηγού απέναντι στις δημόσιες υπηρεσίες και στις απαντήσει που δίνονται στους ευρωπαϊκούς πολίτες. Δύο ερωτήσει έχω να θέσω, θα είμαι σύντομο. Η πρώτη αφορά το, η μέση προθεσμία. Είπατε 66% των ερευνών έκλεισαν μέσα στο έτος. Μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε μια ιδέα για το 44% που μένει, ποια είναι τα περιθώρια προθεσμιών. Και σε ό,τι αφορά το, δίκτυα, το δίκτυο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, τι συμβαίνει των Ευρωπαίων Δημοσιολογητών. Τι συμβαίνει στις χώρες όπου δεν έχετε ε, κάποιο τοπικό συνάδελφο και πώς μπορεί να ενταχθεί κάποιος στο δίκτυο του διαμεσολαβητή στο μέτρο που πολλές ε, ε, αναφορές μπορεί να, να μην απαντηθούν μέσα στα χρονικά όρια που θα κρίνονταν σκόπιμα. Ευχαριστώ. Μποστινάρου. Ευχαριστώ. Κύριε Διαμαντούρο. είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα που παρευρίσκεστε εδώ να μας ε, παρουσιάσετε την έκθεσή σας. Η έκθεσή σας επιβεβαιώνει μια πραγματικότητα που εμείς χαιρετίζουμε. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής αποτελεί ένα μέρος των πιο αξιόπιστων οργάνων, των πιο αξιόπιστων θεσμικών οργάνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τους πολίτες και αυτό σε μια στιγμή που οι εθνικοί θεσμοί αλλά και ευρωπαϊκοί θεσμοί αμφισβητούνται. Έτσι λοιπόν, ε, ο δικός σας ε, θεσμός ε, χαίρει και αυτό οφείλεται στη δική σας δραστηριότητα και της ομάδας σας και το χαιρετίζω αυτό. Έχω μια ερώτηση. Πώς σκοπεύετε στο μέλλον να αναπτύξετε τη συνεργασία με τους εθνικούς διαμεσολαβητές και Μπορούμε να πάρουμε σημείο φετηρίας ε, τρεις ε, περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν εδώ στη δική μας Επιτροπή Αναφορών και καλύπτουν ένα μέρος της εθνικής ευθύνης αλλά και της ευρωπαϊκής ευθύνης. Ε, τα αποτελέσματα του ε, βουλγάρου συνηγόρου του πολίτη, επίσης τα αποτελέσματα του ρουμάνου συνηγόρου του πολίτη και εδώ με την Πρόεδρο αξιολογήσαμε πάρα πολύ καλά τα αποτελέσματα αυτά. Και επίση έχουμε και τη δραστηριότητα του Πολωνού διαμεσολαβητή συνεγόρου του πολίτη, αν θέλετε, ο οποίος προσωπικά δεσμεύτηκε και επέδειξε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Τι θα πράξετε εσείς έτσι ώστε αυτή η υπεραξία που προέρχεται από τη δραστηριότητα των εθνικών συνηγόρων του πολίτη να μεταφραστεί σε κοινού κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και συμπερασματικά να πω ότι προφανώς ε, επένους μόνο έχουμε να σας απευθύνουμε, όμως πιστεύω ότι τα μέτρα λιτότητας ε, δεν μπορούν να αποτελούν μια καθολική λύση. Ξέρουμε ότι το πιο αποτελεσματικό σύστημα είναι ένα δικτατορικό σύστημα και ένα τέτοιο σύστημα ε, μπορεί να μας προφυλάσσει από κάθε δαπάνη. Όμως ε, ο Ευρωπαϊο Δημοσιολαβική χρειάζεται τη χρηματοδότηση ως θεσμό και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι λογικό για να δώσει σε ένα τέτοιο ευρωπαϊκό θεσμό του απαραίτητου πόρου. Καθώς τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ σημαντικά για τους πολίτες. Καλό κουράγιο για τη συνέχιση του έργου σας. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρο. ευχαριστώ. Δεν ζητά άλλο το λόγο. Έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω γενικά ότι θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη που έλαβαν το λόγο, να ευχαριστήσω επίσης την Επιτροπή ε, για ε, τα εγκόμια που μου απίθυναν και είμαι ευγνώμων διότι αυτό αυξάνει το αίσθημα υπευθυνότητας που έχω απέναντι σε αυτό το όργανο και απέναντι στους πολίτες ε, και έτσι αυξάνεται ο πύχης για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους πολίτες και τα όργανα. Θα ήθελα να απαντήσω σύντομα στις ερωτήσεις σχετικά με τις παρατηρήσεις του κ. Νίμαν Κρίστενσεν. Τον ευχαριστώ ε, για τα εγκομιαστικά του λόγια και θα ήθελα να πω ότι δύο ε, τρίτα ε, είναι της, των υπηρεσιών είναι στην Κομισιόν και ελπίζω ότι το ποσοστό αυτό θα βελτιωθεί και βασίζομαι στη συνεργασία σας. Χαίρομαι που οι αρχές των δημοσίων υπηρεσιών που έθεσα είναι κάτι από το οποίο μπορείτε να επωφεληθείτε και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στην Κομισιό. Είναι ακριβώς ο στόχος μου για να υπάρχει ένας οδηγός, ένας οδηγός μίας σελίδας που θα είναι εύκολο να το διαβάσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι όταν έχουν καθημερινά ηθικά διλήμματα και νομίζω έτσι θα μπορέσουν να βελτιώσουν την εργασία τους και χαίρομαι που το εκλαμβάνετε με αυτόν τον τρόπο και υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω στο δρόμο αυτό. Σας ευχαριστώ και πάλι. Κυρία Σινκλέρ, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Εκτιμώ την ειλικρίνεια και ευθύτητα και θα πάρω τα πράγματα με τη σειρά τους. Η πρώτη κατηγορία με τον κατάλογο των χωρών γεωγραφικά αναφέρεται σε δύο κατηγορίες. Πρώτον, η κατηγορία των προσφυγών που προέρχονται από χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δεύτερη αναφέρεται σε προσφυγές που ήρθανε ε, χωρίς προέλευση, χωρίς αναφορά προέλευσης. Και, και αυτό, ε, με αυτά τα δύο κατηγορίες έχουμε το άθροισμα θα πρέπει να σας πω ότι επιφυλακτικά συμφωνώ μαζί σας ως προς το θέμα ότι ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής δεν είναι αρκετά γνωστός στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν είναι αρκετά ορατός. Με ρωτάτε τι κάνω, τι πρέπει να κάνω. Κάτι που έχω κάνει κατά τη διάρκεια των ετών, είχα επαφές με την ε, Επιτροπή, την Κοινοβουλευτική των Υπηρεσιών Υγείας και η κυρία Έιμπραχαμ, ήταν ε, θεαματικά επιτυχημένη ε, διαμεσολαβήτρια στην χώρα σας και άφησε μεγάλη κληρονομιά και ελπίζω να μπορέσει να υπάρξει και αλλού μια τέτοια κληρονομιά και ότι ο διάδοχός της θα συνεχίσει το έργο της. Ε, Ρεγάστηκα στενά με την κυρία Ήμπραχαμ, επισκέφθηκα επανειλημμένα το Ηνωμένο Βασίλειο και έλαβα μέρος ε, στην Ένωση των Διαμεσολαβητών Αγγλίας και Ιρλανδίας που είναι ε, το πιο πυκνό δίκτυο διαμεσολαβητών στον κόσμο και μπορώ να σας πω ότι τόσο από την άποψη του αριθμού των επισκέψεων αλλά και από την ε, ένταση, των, την ποιότητα των επισκέψεων μπόρεσα να στιάσω την προσοχή μου στη χώρα σας και μπόρεσα να διατηρήσω το επίπεδο υποστήριξης εκεί κυρίως ε, διαμέσου ε, του, της υποστήριξης του διαμεσολαβητού του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν ξέρω κυρία Σενκλέρ πώς θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τους ευρωβουλευτές για να προωθήσω ε, την εικόνα, την, το ρόλο του διαμεσολαβητού στις χώρες. Δεν χρησιμοποιώ τους ευρωβουλευτές αλλά είμαι στην διάθεση όλων ε, των χωρών. Αν θέλει κανεί ε, από τους Ευρωβουλευτές του Ηνωμένου Βασιλείου να κάνει χρήση των υπηρεσιών μου ε, για να εξοικειώσει τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου για την αποστολή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβήτη σχετικά με τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ τον κύριο Σαλαβράκο και τον κύριο Μποστονάρο που πρόλαβαν κατά κάποιο τρόπο την αντίδρασή μου θα ήθελα να σας πω το εξής. Ο εύκολος τρόπος προσέγγισης του θέματος του προϋπολογισμού είναι να πάρει κανείς τον αριθμό των προσφυγών που έχουν ληφθεί και μετά να διαιρέσει τον προϋπολογισμό δια του αριθμού αυτού. Θα ήθελα όμως να επιστήσω την προσοχή σας ότι εκτός από τα όσα ανέφερα για αυτό το έτος μπορέσαμε να βοηθήσουμε πάνω από 22.000 άτομα με κάποιο τρόπο. Αν λοιπόν ε, διαιρέστε δια του αριθμού των 22.000 υπάρχει μεγάλη μείωση του αριθμού που προκύπτει. Θα ήθελα επίσης να πω ότι χαίρομαι και είμαι ευτυχής που μπόρεσα να ε, αντιδράσω εδώ στις, ε, τα αιτήματα αυτής της Επιτροπής και της Ευρωβουλής ε, και να μειώσω ε, τον αριθμό των απαράδεκτων ε, αναφορών και των προσφυγών και μπορέσαμε να μειώσουμε με τον οδηγό κατά 25%. Ο χαμηλός αριθμός που έχετε είναι απόρρια μιας επιτυχίας, ούτως ώστε να μειώσουμε τον αριθμό Έλαβα υπόψη πέρσι τις παρατηρήσεις σας για τη λιτότητα και θέλω να σας πω τρία πράγματα. Πρώτον, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών είχε τρει διαδοχικούς προϋπολογισμούς όπου η αύξηση δεν ξεπέρασε το 0,1%. Ε, είχαμε 0,10 έως 0,14, 0,15 Συνεπώς νομίζω ότι υπάρχει απτή απόδειξη ότι ο διαμεσολαβητής έχει πλήρη συνείδηση της ανάγκης ε, τήρησης της αρχής της λιτότητας για την ώρα. Ο λόγος ε, του ύψους για φέτος ε, σας δόθηκε από τους συναδέλφους σας. Το Κοινοβούλιο στη σοφροσύνη του αποφάσισε να μετακομίσει ο διαμεσολαβητής για να χρησιμοποιηθούν ε, τα γραφεία για το Μουσείο Ιστορίας της Ευρώπης. Ε, μετακομίζουμε λοιπόν σε νέα γραφεία και έχουμε σημαντικά έξοδα. Έχουμε ενίκιο σημαντικό το οποίο ε, για το κτίριο Eastman και λοιπόν έχουμε ένα, ένα πρόσθετο έξοδο που οφείλεται στο Κοινοβούλιο ιστορικά. Το Κοινοβούλιο βοηθάει τον διαμεσολαβητή ε, παρέχοντας του ένα λογιστή που λαμβάνει υπόψη τα οικονομικά μας. Ενημερωθήκαμε ότι ο λογιστής θα αποσπαστεί αλλού, θα αναλάβει άλλες ευθύνες και συνεπώς έχουμε υποχρέωση ε, να έχουμε έναν λογιστή που να αναλάβει την εργασία αυτή βάσει του οικονομικού κανονισμού. Γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε να πληρωθεί αυτή η θέση. Ελπίζω να απήντησα σε όλα τα θέματα τα οποία σας απασχολούν. Κύριε Άουτγκαν, σας ευχαριστώ και πάλι για τις παρατηρήσεις σας και για την υποστήριξη στο έργο του διαμεσολαβητού. Είμαστε ευγνώμονες. Θα ήθελα να επαναλάβω τα όσα είπατε, ότι πώς κάποιος ερμηνεύει τον υψηλό αριθμό προσφυγών. Η ερμηνεία αυτή μπορεί να ποικίλει πάρα πολύ βεβαίως. Δεν νομίζω ότι ο υψηλός αριθμός προσφυγών είναι ένδειξη προβλήματος. Το γεγονός ότι έχετε σε απόλυτους αριθμούς τον μεγαλύτερο αριθμό προσφυγών που να προέρχεται από την Ισπανία που είναι ε, μικρότερη χώρα από την Γερμανία και μπορώ να σας πω ότι στα 5-6 τελευταία χρόνια η Ισπανία είχε δύο-τρεις περιπτώσεις όπου ξεπέρασε την Γερμανία σε απόλυτους αριθμούς. Αυτό ε, δεν δείχνει βέβαια ότι οι Ισπανοί μονίμως παραπονούνται, αλλά ότι έχουν ότι έχουν μια σειρά θεσμών στη χώρα τους, όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Σημερίζουμε λοιπόν την παρατήρησή σας και σας ευχαριστώ που την αναφέρετε σχετικά με το διοικητικό δίκαιο ε, το ευρωπαϊκό. Ξέρετε ποια είναι η θέση του διαμεσολαβητή. Η ευθύνη μου και η αποστολή μου είναι να εφαρμόζω αυτό που αποφασίζει αυτό το αξιότιμο σώμα. Όταν υπάρχει νομοθεσία, εγώ ε, την υλοποιώ, την εφαρμόζω. Εάν ο νομοθέτης ο Ευρωπαίος υιοθετήσει ε, δίκαιο διοικητικό θα το εφαρμόσουμε και θα το εφαρμόσουμε με τον ίδιο τρόπο όπως γίνεται τώρα. Θα εξετάσουμε τον νόμο όσο το ελάχιστο προαπαιτούμενο για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι άνθρωποι και επιπλέον θα εφαρμόσουμε τις αρχές της κακής διοίκησης που εξορισμού είναι κάτι το ευρύτερο από τον νόμο. Περιμένω λοιπόν τις αποφάσεις του νομοθέτη ως προς το θέμα αυτό. Τέλος, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σας ότι δεν είναι μόνο οι πολίτες αλλά και η δίκηση που έχουν σημασία και που θα ωφεληθούν από τέτοιου είδους κανονισμό. Ε, κύριε Σαλαβράκο, θα ήθελα να σας απαντήσω στην ε, κοινή μας γλώσσα, αν μου το επιτρέπετε. Πάρα πολύ κύριε Σαλαβράκο που με κρίνεται με αυστηρότητα. Διότι αυτό περιμένω από τα μέλη του Κοινοβουλίου, ενώπιον των οποίων εμφανίζομαι προκειμένου να εξηγήσω και να παρουσιάσω τις ειδήσεις εκθέσεις μου και δεν θα περίμενα τίποτα λιγότερο από σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω εγώ τα, τα σχόλια εκείνα τα δικά σας τα οποία αφορούν την τρέχουσα πολιτική συγκυρία για την οποία ως Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής δεν θα έπρεπε να πάρω θέση. Ε, απλώς να πω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι το αίσθημα δικαιοσύνης είναι ευρύτερο του ε, αισθήματος απονομής δικαιοσύνης και ότι αυτό κατά κάποιο τρόπο λειτουργεί παράλληλα με την διάκριση που κάνει πάνω ο διαμεσολαβητής μεταξύ νομιμότητας και χρηστής διοίκησης. Και πάλι σας ευχαριστώ και για τα σχόλιά σας και για την διευκρίνηση σε ό,τι αφορά το θέμα του προπολογισμού μου που είχατε την καλοσύνη να κάνετε ε, σχολιάζοντας τα σχόλια της κυρίας Συγκλέα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπουλόν για τις παρατηρήσεις σας και επιτρέψατε μου να απαντήσω με τη σειρά, ακολουθώντας τη σειρά των ερωτήσεών σας σχετικά με το χρόνο, την προθεσμία που χρειαζόμαστε για να κλείσουμε ορισμένες ε, περιπτώσεις και υποθέσεις, μπορώ να σας πω ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αρκετά ικανοποιητική, διότι τα τρία τελευταία χρόνια μπορέσαμε να μειώσουμε το μέσο όρο του χρόνου που απαιτείται για να κλείσουμε ορισμένες ε, υποθέσεις και τώρα ο μέσος όρος είναι περίπου 9 μήνες. Τούτων λεχθέντων εποφελούμε από την ευκαιρία αυτή για να σας αναφέρω ότι στην δεκαετία του 60 του περασμένου αιώνα υπήρξε ένα βιβλίο αρκετά γνωστό του οποίου ε, τίτλος είναι «Πώς να λέει κανείς ψέματα με τις στατιστικές». Θα πρέπει λοιπόν να είμαι διαφανής ως διαμεσολαβητές και σας είπα ότι ο μέσος όρος δείχνει ότι σε περιπτώσεις που μπορούμε να κλείσουμε υποθέσεις είναι τρεις μήνες, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις περίπλοκες όπου ξεπερνάμε το χρόνο και χρειαζόμαστε και 1,5 χρόνο. Ο μέσος όρος είναι 9 μήνες. Πέραν λοιπόν από το 55% των υποθέσεων κλείνουν πριν το τέλος ενός έτους και μπορέσαμε να μειώνουμε, μπορούμε να μειώνουμε συνεχώς την, τον χρόνο από το 2008 που εισαγάγαμε νέες διαδικασίες που μας επιτρέπουν να επιταχύνουμε τον τρόπο διεκπαιρέωσης και αντιμετώπισης των προσφυγών. Η δεύτερη σας ερώτηση, πώς προσπαθώ να προωθήσω τις σχέσεις όπου δεν υπάρχουν σε χώρες διαμεσολαβητές. Ο διαμεσολαβητής υπάρχει μόνο στην Ιταλία σε επίπεδο εθνικό. Στη Γερμανία υπάρχουν οι επιτροπές αναφορών που υπάρχουν είτε ε, στο επίπεδο της Ομοσπονδίας είτε στο επίπεδο των κρατηδίων και υπάρχουν τέσσερις ή πέντε ε, Διαμεσολαβητέ στο επίπεδο των Λέντερ, των κρατηδίων. Εκεί υπάρχει μια άλλη διευθέτηση που μας επιτρέπει μια άμεση σχέση, μια άμεση επαφή με τους Γερμανούς συναδέλφους. Στην Ιταλία δυστυχώς το πρόβλημα είναι σοβαρότερο διότι σε εθνικό επίπεδο η Ιταλία είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει ε, μη δικαιοδοτικά μέσα προσφυγής επεσκέφθη την Ιταλία πάνω από δέκα φορές προσπαθώντας να προωθήσω μια τέτοια ενδεχόμενη οθέτηση ενός νόμου. Ε, δύο χρόνια ε, συζητώ με τον πρόεδρο Ναπολιτών και σύμφωνα με τις πληροφορίες μου ίσως η σημερινή κυβέρνηση να είναι πιο διατεθειμένη να εξετάσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο και είμαι πάντοτε στη διάθεσή τους και έστειλα σημειώματα και ενδείξεις ότι είμαι διατεθειμένος να πάω και πάλι στην Ρώμη για να βοηθήσω σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Στην Ιταλία, ξέρετε βεβαίως, νομίζω ότι το τοπικό επίπεδο εξαλείφθηκε πλήρως πέρσι ε, για την διαμεσολάβηση και υπάρχει μόνο σε επίπεδο περιφερειακό. Υπάρχουν 20 περιφέρειες στην Ιταλία και μόνο 11 από αυτές έχουν περιφερειακούς ε, διαμεσολαβητές. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο κενό στην Ιταλία και είμαι πάντοτε έτοιμος να βοηθήσω κάθε προσπάθεια για την βελτίωση της κατάστασης. Κύριε Μποστινάρο, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, γιατί λόγω τεχνικών προβλημάτων έχασα την αρχική, το αρχικό ε, σημείο της παρέμβασής σας, αλλά δεν έχασα τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ για το τμήμα που άκουσα <coughs> σχετικά με την υψηλή σας εκτίμηση για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και για όλα τα εγκόμια, όπως είπα, αυξάνουν το αίσθημα ευθύνης μας για να κάνουμε την εργασία μας με ε, ικανοποιητικό τρόπο. Σε σχέση με τις ερωτήσεις... do Τι συμβαίνει ούτως ώστε ο εθνικός διαμεσολαβητής να μπορεί να προωθήσει μια κατάσταση. Το βασικό μέσο που έχουμε είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών. Αν το χρησιμοποιούμε καλά το σύστημα αυτό για ανταλλαγέ πληροφοριών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, για να μπορούμε να λαμβάνουμε προσφυγές από τους εθνικούς ομολόγους μας και να του στέλνουμε προσφυγές, επιπλέον λαμβάνουμε έρευνες, ε, αιτήματα για έρευνες από εθνικούς συναδέλφους σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πάρα πολλές τρόποι συνεργασίας για να μπορέσουμε να επιτύχουμε δύο στόχους. Να αυξήσουμε την γνώση που υπάρχει στα κράτη-μέλη για το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι ξέρουμε ότι πρόκειται για μια καθημερινή πραγματικότητα στα κράτη-μέλη, γι' αυτό θα πρέπει να γίνει αυτό κατανοητό στο βασικό επίπεδο και στο επίπεδο των δημοσίων υπηρεσιών, όπου η Εθνική συνάδελφοι μπορούν να τους ενημερώσουν και στο επίπεδο το δικαστικό, πράγμα που κάνω εγώ, τους ενημερώνω όταν επισκέπτομαι τα κράτη-μέλη. Αναφέρατε τη χώρα σας, αναφέρατε τη Βουλγαρία, νομίζω ότι η Βουλγαρία τώρα έχει έναν εξαιρετικό νέο διαμεσολαβητή με τον οποίο ε, συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά και προσπαθούμε να αναδιαρθρώσουμε την υπηρεσία του για να μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα τους συμπατριώτες του στην αρχή του 2013. Έχω δεσμευθεί απέναντι στον κύριο Γιάνκο ότι θα επισκεφθώ τη χώρα σας και θα επωφεληθώ του γεγονότος ότι ο κύριος Γιάνκο είναι ο καινούριο διαμεσολαβητής της χώρας και ήταν πάρα πολύ δραστήριος για να έχει αναλάβει νέες πρωτοβουλίες ούτω ώστε το όργανο αυτό να γίνει καλύτερα γνωστό στους πολίτες και πάλι ε, σας ευχαριστώ και εσάς και τον κύριο Σαλαβράκο ε, για τα σχόλιά σας ε, σχετικά με τον προϋπολογισμό μου. Το μόνο που μπορώ να πω είναι αυτό που είπα στην κυρία Σενκλέρ ότι η αύξηση του προϋπολογισμού κατά κάποιο τρόπο οφείλεται στο Κοινοβούλιο. Δεν τη ζητήσαμε εμείς αυτή την αύξηση. Τα τελευταία χρόνια ζητήσαμε αυξήσεις που ήταν κοντά στο μηδέν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Διαμαντούρο για την παρέμβασή του και ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη συζήτηση και σίγουρα οι ιδέες ε, που ακούστηκαν ε, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ε, και για την έκθεση που έχω να καταρτήσω εγώ για την επόμενη συνεδρία του Ιουλίου κατά την οποία θα συζητήσουμε και εμείς ως Επιτροπή εις βάθος ε, τους προβληματισμούς που ακούστηκαν σήμερα. Όμως ε, δεν θα απελευθερώσουμε το λαβητή γιατί στο επόμενο σημείο έχουμε και πάλι παρέμβασή σας να μας παρουσιάσετε την ειδική έκθεση σχετικά με την έρευνα, σχετικά με την καταγγελία 2591 του 2010 την προσφυγή 2591-2010 κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει ως αντικείμενο την επέκταση του αεροδρομίου της Γέννης. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Διαμαντούρο για να μας παρουσιάσει το σημείο αυτό. <clears throat> All right. Thank you again. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ξανά που μου δώσατε το λόγο δεύτερη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να κάνω μια σύντομη παρουσίαση βασισμένη στην συμφωνία μας ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής θα οφείλει να παρουσιάζεται ενώπιόν σας όποτε υποβάλλει μια ειδική έκθεση στο Κοινοβούλιο. Οι ειδικέ εκθέσεις είναι το ε, το όπλο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Όπω παρουσίασα και πριν στην ετήσια έκθεση, οι αποφάσει μου δεν είναι νομικά δεσμευτικέ. Επομένω, λοιπόν, εξαρτώμαι στην ικανότητα που έχω να σας πείσω με επιχειρήματα και επίσης στην δύναμη της κοινή γνώμης και της δημοσιότητας έτσι ώστε να επιτύχω την συμμόρφωση με τι συστάσεις που δίνω. Ο πολύ μικρός ε, αριθμό ειδικών εκθέσεων που έχει παρουσιάσει ο διαμεσολαβητής στο Κοινοβούλιο, 18 σε 16,5 ε, χρόνια, πιστεύω ότι αποτελεί απόδειξη της ε, προσέγγισης που έχει οθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πλειοψηφία των υποθέσεων. Ένα... Υπάρχει όμως η γνώση ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής έχει τη δυνατότητα να κάνει μια ειδική έκθεση και ιδιαίτερα όταν γίνεται ένα σχέδιο για σύσταση γνωρίζουμε ότι το επόμενο, γνωρίζοντας ότι το επόμενο βήμα θα είναι μια ειδική έκθεση ασκείται πίεση για, ε, για να αλλάξει την στάση του η, τη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εδώ το Κοινοβούλιο έχει έναν τρόπο για να πείσει λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως πολιτικό όργανο συνδέεται με τις ειδικέ εκθέσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Ελπίζω ότι όταν εξετάσει μια ειδική έκθεση, το Κοινοβούλιο πάντα θα λαμβάνει υπόψη του ότι το δικαίωμα των αιτήσεων είναι θεμελιώδες δικαίωμα ενός Ευρωπαίου πολίτη, ότι υπάρχει στην Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που με τη συνθήκη της Λισαβόνας είναι νομικά δεσμευτική. Για τους λόγους που ανέφερα ήδη, οι ειδικέ εκθέσεις στο Κοινοβούλιο και οι απαντήσεις σε αυτές αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του έργου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Τώρα θα προχωρήσω στην ειδική έκθεση που παρουσίασα στις 14 Μαΐου στο Κοινοβούλιο για την υπόθεση 2591 του 2010 με αρχικά GG. Πιστεύω ότι συνοπτικά η Κομισιόν έχει αποτύχει να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι οι Αυστριακές αρχές αναμίχθηκαν σε μία σύγκρουση συμφερόντων στην διαχείριση του ζητήματος αυτού, ότι υπήρξε έλλειψη ε, διαδικασιών ε, ε, εξέτασης στις προσφύγες αυτές. Θέλω την βοήθεια του Κοινοβουλίου έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι η διαδικασία αυτή αναθεώρησης θα είναι δυνατή. Η υπόθεση αυτή αναφέρεται στην επέκταση του αεροδρομίου της Βιέννης με πολλά νέα κτίρια με την άδεια των Αυστριακών Αρχών. Σύμφωνα με, την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να κάνουν μία ε, EIA, μία περιβαλλοντική εκτίμηση αντικτύπου. Το 2006 υπήρξαν 27 πρωτοβουλίες πολιτών για τις αρνητικές συνέπειες ε, του, της επέκτασης του αεροδρομίου της Βιέννης και διατύπωσαν προσφυγή στην Κομισιόν λέγοντας ότι αυτές οι, περιβαλλοντικές εκτιμήσεις αντικτύπου δεν διεξήχθησαν από τις αυστριακές αρχές. Όμως, από τότε που τα σχέδια επέκτασης, όμως καθώς τα σχέδια επέκτασης είχαν σχεδόν ολοκληρωθεί, συμφωνήθηκε με τις αφριστριακές αρχές ότι δεν θα συνεχίζονταν οι διαδικασίες για την παράβαση και ότι θα, μάλλον ότι θα απέφευγαν να συνεχίσουν την, ε, τις έρευνες για τη διαδικασία παράβασης. υπήρξε δυσαρέσκεια με τον τρόπο που οι αυστριακές αρχές έκαναν την εκ των υστέρων περιβαλλοντική εκτίμηση αντικτύπου. Η αρχή που της είχε ανατεθεί η εκτίμηση αντικτύπου αυτή ήταν η ίδια αρχή που είχε ορισμένες άδειε εκτέλεσης των έργων επέκτασης. Και αυτό δεν συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Το αρμόδιο Υπουργείο που είχε εκδώσει ορισμένες άδειες ήταν επίσης αναμεμειγμένο στην υπόθεση αυτή. Και κατόπιν εξέτασης της υπόθεσης συμμερίζομαι την άποψη των καταγγελόντων. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε δώσει, δεν είχε απαιτήσει μάλλον εγγυήσεις από την Αυστριακή κυβέρνηση ότι έχουν γίνει αυτές οι περιβαλλοντικές εκτιμήσεις αντικτύπου, τα EIAs. Συμπεραίνω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διασφάλισε την ε, διεξαγωγή και την κατάλληλη μάλιστα διεξαγωγή των εκτιμήσεων αντικτύπου. Η Κομισιόν είχε δηλώσει ότι η υπόθεση θα έκλεινε μόνο όταν Υπήρχε διαβεβαίωση ότι οι αυστηριακέ αρχέ είχαν λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Γι' αυτό λοιπόν θεώρησα ότι δεν υπήρχε ανάγκη για περαιτέρω ε, σε εκείνο το στάδιο και είχα εμπιστευτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα λάμβανε υπόψη την συστάσει μου. Το 2010 οι καταγγέλλοντες απευθύνθηκαν πάλι σε μένα και ισχυρίστηκαν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε κάνει κανένα παραπάνω βήμα ε, και δεν είχε κινήσει καμία διαδικασία εναντίον της Αυστρίας. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισα να αρχίσω δεύτερη έρευνα, δεύτερη διαδικασία για το ζήτημα αυτό. Συνέταξα ένα σχέδιο σύστασης το 2011 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξετάζοντας το ντοσιέ είδα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όντως δεν είχε λάβει περαιτέρω δράσεις για τα ζητήματα τα οποία της είχα επιστήσει. Δεν υπήρχε τίποτα στον φάκελο που αποδείκνυε ότι η Κομισιόν είχε συζητήσει γραπτός με τις Αυστριακές Αρχές το ζήτημα αυτό. είχε ολοκληρωθεί η πρώτη διαδικασία παραβάσεις επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με είχε διαβεβαιώσει ότι θα έκλεινε την υπόθεση μόνο όταν είχε ικανοποιητικές αποδείξεις ότι οι αυστριακές αρχές είχαν αντιμετωπίσει και εξετάσει το ζήτημα. Και θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπρεπε να είχε λάβει υπόψη τις συστάσεις που είχα δώσει στην πρώτη σύσταση. Ειδικά ω ό,τι αφορούσε την σύγκρουση συμφερόντων, γιατί πιστεύω ότι υπήρχαν βάσιμες αποδείξεις για σύγκρουση συμφερόντων. Έγινε μετά τον έλεγχο από το Συμπαράλληλα, λοιπόν, ότι και μετά από, τις, ε, από την εξέταση του ελεκτικού συνεδρίου της Αυστρίας, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έλαβε σοβαρά υπόψη της συστάσεις μου. Η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο σχέδιο της σύστασης δεν αντικατόπτριζε τις απόψεις μου ούτε στην πρώτη ούτε κατά την δεύτερη σύσταση σε ό,τι αφορά την σύγκρουση συμφερόντων και την εξέταση περιβαλλοντικού αντικτύπου. Ούτε έλαβε υπόψη τις ανησυχίες των πολιτών. Αντίθετα, μάλιστα, φάνηκε ότι είτε δεν θεώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγκαίο να καθορίσει εάν γίνεται να υπάρξει διαδικασία αναθεώρησης για εκ των υστέρων ε, εκτίμηση περιβαλλοντικού αντικτύπου, είτε να πείσει τους ε, καταγγέλλοντες και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ότι μια τέτοια διαδικασία δεν ήταν απαραίτητη διότι δεν ίσχυαν οι κατηγορίες αυτές. Και αυτό ε, μας δίνει ενδείξεις για μη σωστή δίκηση, για αποτυχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξετάσει την σύγκρουση συμφερόντων και την νομιμότητα του έργου αυτού. Εάν θυμάμαι καλά, οι αυστριακές αρχές είχαν εκδώσει άδεια εργασιών χωρίς να έχουν κάνει περιβαλλοντική εκτίμηση αντικτύπου. Γι' αυτό λοιπόν δεν ήταν πεπισμένες οι αυστριακές αρχές. Θα ήθελα να ζητήσω από το Κοινοβούλιο να ζητήσει με τη σειρά του από την Επιτροπή να αναθεωρήσει τη θέση της για την διαχείριση του, της προσφυγής αυτής των πολιτών της Αυστρίας για την επέκταση του αεροδρομίου της Βιέννης. Αυτό σημαίνει ότι οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να λάβουν υπόψη την υποχρέωση των εθνικών αρχών να διασφαλίσουν ότι καταρχάς οι καταγγέλλοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβαση σε διαδικασία αναθεώρησης και δεύτερον ότι τα κατάλληλα βήματα θα ληφθούν για να εφαρμοστεί η Οδηγία 85 κάθετος 337. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Διαμαντούρο. Το λόγο έχει τώρα ο πρόσωπος της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι γενικά υπήρξε μια καλή συνεργασία μεταξύ της ε, Κομισιόν και του Διομεσολαβητή σε περιβαλλοντικά θέματα. Ένα παράδειγμα είναι στην ανακοίνωσή μας για την εφαρμογή. Λάβαμε κάποιες ιδέες από το Διομεσολαβητή σε σχέση με το δίκτυο των διαμεσολαβητών. Λέχθεντος αυτού, φοβάμαι ότι ξεκολουθούμε να διαφωνούμε μεταξύ μας και ξεκολουθούμε να έχουμε και κάποια ερωτηματικά σχετικά με την έκθεση που εκπονήσατε, την οποία βέβαια τη λαμβάνουμε πολύ σοβαρά, γιατί δεν ξεκίνησε κάποια διαδικασία σε αυτό το οίκο. Θα ήθελα να αναφέρω τι ζητήματα έχουμε. Έχουμε δύο μεγάλες συζητήσεις ε, που λαμβάνουν χώρα Καταρχήν, ε, σε σχέση με το ποιο είναι ο στόχο μια διαδικασία επιπαραβάση, όταν ε, η παραβίαση, η παράβαση αυτή έχει γίνει πριν πολλά χρόνια. Και το δεύτερο ζήτημα, η δεύτερη ομάδα ζητημάτων είναι ποια είναι η διαφορά μεταξύ των νομικών υποχρεώσεων δυνάμει τη οδηγία ε, μελέτη αντικτύπου, που μπορεί να επιβάλλει κομισιόν και τι θα μπορούσε να είναι από τη δίκηση των κρατών μελών. Αυτά θα ήθελα να τα τονίσω. Για το πρώτο ζήτημα Μιλάμε για ένα μικρό έργο, όπως παραδείγματος χάρη, ένα πύργο ανακαίνιση των συστημάτων φωτισμού που άρχισαν να εφαρμόζεται το 1999 και λάβαμε γι' αυτά προσφυγή το 2006. Έτσι είχε η κατάσταση που αντιμετωπίσαμε και οι καταγγέλλοντες θα μπορούσαν να προσφυγούν στο Αυστριακό Δικαστήριο και Πράγματι, άλλοι καταγγέλλοντε ε, κατά τι επέκταση αυτού του προσέφηκαν στο δικαστήριο και τώρα εκκρεμούν υποθέσει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. C420-11 είναι η υπόθεση. Έτσι λοιπόν, ε, το δικαστήριο θα αποφανθεί. Βρισκόμαστε λοιπόν στην κατάσταση όπου χτίστηκαν κάποια κτίρια κατά παραβίαση της οδηγίας πριν μελέτης αντικτύπου. Και τι κάνουμε. Βασικά έχουμε δύο επιλογές, δύο εναλλακτικέ. Η μία είναι να προσπαθήσουμε να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερα μέτρα αντιστάθμισης αποζημίωσης από τις αρχές, ενώ η άλλη λύση είναι πράγματι να προσφύγουμε στο δικαστήριο, να προσπαθήσουμε να κυρώσουμε την άδεια και να καταστραφεί η επένδυση. Αυτή είναι μια διαδικασία, ένα αποτέλεσμα της διαδικασίας επί Φαίνεται ακραίο στην κατάσταση. Αυτή είναι ακραία η κατάσταση, αλλά την ε, μάθαμε ότι κάτι τέτοιο το σκεφτόμαστε σε μια χώρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης κατά ενός υλικού πάρκου. Είναι μια ακραία επιλογή, αλλά υπάρχει λοιπόν. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε, ας χρησιμοποιήσουμε τη διαδικασία επί παραβάση και ας προσπαθήσουμε να έχουμε δυνατόν περισσότερες αποζημιώσεις από τις αυστριακές αρχές και δεν νομίζω ότι διαφωνούμε κύριε Διαμεσολαβήτη σε αυτό. Θέλουμε να έχουμε μία μελέτη αντικτύπου ex post, ε, λαμβάνοντα υπόψη ότι δεν μπορεί να διορθωθεί πλέον η κατάσταση. Και μάλλον εδώ θα ξεκινήσει η διαφωνία μα. Νομίζω ότι είμαστε, ασκήσατε κριτική για το γεγονό ότι δεν ε, κάναμε αρκετά για να ελέγξουμε αυτή την ex post μελέτη αντικτύπου, περιβαλλοντική μελέτη αντικτύπου. Πιστεύουμε ότι η νομοθεσία ω έχει δεν μα επέτρεψε να πάμε παραπέρα σε ό,τι φορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Όπως ε, αναφέρεται στην παράγραφο 53 της εκθεσής σας, ε, θα ήταν ε, δίκαιο θεμητό να υπάρχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη, όμως αυτό δεν αρκεί για μας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους κανόνες του αστικού κώδικα ή του κώδικα διαδικασίας. Χρειαζόμαστε παράβαση και η Αυστρία δεν θα μπορούσε να παρακάμψει του κανόνε της ε, για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, για αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση. Έτσι λοιπόν ε, πιστέψαμε ότι δεν μπορούσαμε να πάμε παραπέρα για το σημείο αυτό. Σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων, ε, η οδηγία μελέτη αντικτύπου δεν ρυθμίζει κάτι τέτοιο. Είναι κρίμα. Είναι δυνατό, αλλά αν το δείτε, αν το σκεφτείτε μάλλον, όταν ένα δικαστήριο ή ένας ε, ανώτερος ε, φορέας καταργήσει μια άδεια, θα στείλει την απόφαση πίσω σε αυτή την αρχή. Ακόμη και αν ε, το δικαστήριο ακυρώσει μια απόφαση ενός περιφερειακού δικαστηρίου, θα το στείλει πίσω στο περιφερειακό δικαστήριο και δεν θα θεωρηθεί ότι υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων. Έτσι λοιπόν δεν θεωρώ ότι είναι βέλτιστη η κατάσταση αυτή, όμως κατά τη δική μας ερμηνεία της οδηγίας της μελέτης αντικτύπου, τίποτα περισσότερο δεν μπορούσαμε να κάνουμε παρά να επισημάνουμε το θέμα αυτό στις αρχές. Και σας διαβεβαιώ ότι τη δική σας έκθεση τη διαβιβάσαμε στις αρχές της Αυστρίας και τη συζητήσαμε, αλλά τίποτα δεν μπορούσε περαιτέρω να βγει από τη διαδικασία επί παραβάση. Και κάτι που θέλω να αποσαφηνίσω γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντικό για το μέλλον. Στην παράγραφο 57 αμφισβητείται το γεγονός ότι εκμεταλλευόμαστε τη νέα περιβαλλοντική μελέτη αντικτύπου και την επέκταση του αεροδρομίου και λέτε πώς μπορεί να υπάρχει κάποια διστάθμιση. Τώρα, η σημερινή μελέτη δικτύπου που συνεχίζεται θα υπολογίσει το σωρευτικό αντίκτυπο των δύο έργων, των δύο project. Έτσι λοιπόν, για το σημείο αυτό, Πρέπει να δούμε τι θα σημαίνει αυτή η νέα μελέτη αντικτύπου. Από νομική σκοπιά θα έχουμε μια σωρευτική αξιολόγηση του προηγούμενου project με τον ίδιο τρόπο. Αν θέλουμε δηλαδή νέα άδεια για ανεμογεννήτρες κάπου στην Ρουμανία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις υφιστάμενες ολογεννήτριε. Έτσι λοιπόν από νομική σκοπιά οι αυστριακέ αρχέ υποχρεούνται να κάνουν κάτι τέτοιο και εξακολουθούμε να είμαστε σε επαφή με τις αυστριακές αρχές και έχουμε επιβεβαίωση ότι η δική τους μελέτη αντικτύπου λαμβάνει πλήρως υπόψη τον αντίκτυπο των προηγούμενων έργων. Τώρα η κύρια πρόκληση για αυτό το αεροδρόμιο είναι ο θόρυβος. Αυτό είναι ο μεγαλύτερο αντίκτυπο για του πολίτε και έχουμε πληροφορίε. Μπορούμε να μοιραστούμε με τον μελλοντικό συγητή. Πράγματι, οι αυστριακέ αρχέ λαμβάνουν υπόψη σοβαρά τον αντίκτυπο του θορύβου και αν ε, το σκεφτείτε, είναι πιο εύκολο να υπολογίσει κανεί τον αντίκτυπο του θορύβου ενό ε, νέου τρίτου ε, διαδρόμου προσγείωση από ότι ενός χώρου πάρκινγκ. Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση αυτή, οι αυστηριακές αρχές ε, μπορούν να κάνουν ε, τη δουλειά τους καλά, όμως το θέμα είναι ο θόρυβος που θα προκληθεί από αυτή την επέκταση του αεροδρομίου. Πιστεύουμε ότι δικαίω τονίζει τουρισμένα προβλήματα, όμως πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τα όρια του νόμου, μάλλον ε, αποτύχαμε να έρθουμε σε ε, επαρκή επικοινωνία μαζί σας ε, και με τον καταγγέλλοντα, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ποια είναι τα όρια της διαδικασίας επί παραβάση. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ και τον διαμεσολαβητή για την παρέμβασή του. Δεν βλέπω να ζητά κάποιος το λόγο. Κύριο Βαστινάρου, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως ο Σέξπιρ με τις απαντήσεις που λάβαμε σήμερα, αυτές οι απαντήσεις προκαλούν νέες ερωτήσεις. Διότι, πρώτον, η περίπτωση που αναφέρατε κυρία Διαμεσολαβητά είναι για μας μια ιδιαίτερη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί διότι πρόκειται για την αξιοπιστία της αξιολόγησης περιβαλλοντικού αντικτύπου όταν γίνονται από τους επενδυτές αυτές οι αξιολογήσεις. Όπως σε πολλές άλλες περιπτώσεις σε όλη την Ευρώπη πρόκειται για πραγματική σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στον επενδυτή και στην αξιοπιστία των αξιολογήσεων περιβαλλοντικού αντικτύπου. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, αυτό συνέβη στην Αυστρία. Μια, ένα κράτος ε, που έχει μια δημόσια δίκηση εύρωστη, στερεά, ε, ε, στιβαρές εθνικές αρχές, επιβολή νόμου που γίνεται με το σωστό τρόπο. Φανταστείτε αυτό να συνέβαινε σε άλλα κράτη-μέλη όπου οι αρχές Ε, δεν είναι όπως στην Αυστρία, στην Ρουμανία. Έχω, έχω, μπορώ να, μιλήσω για τη Ρουμανία. Μπορούμε να ε, εμπιστευτούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάθε ότι κάθε κράτος μέλος θα ε, εφαρμόζει πλήρως τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Ωραία είναι οι κανόνες, ακόμα και τέλεια, αλλά στην πράξη θέτουν σοβαρό πρόβλημα η υλοποίησή τους και η τελευταία μου ερώτηση, γιατί χρειαζόμαστε τη νέα οδηγία για την αξιολόγηση περιβαλλοντικού αντικτύπου ζητήσαμε επανειλημμένα ότι χρειαζόμαστε μια νέα τέτοια οδηγία ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα από την το σωρευτικό αντίκτυπο και έρχομαι στη δική μου περίπτωση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας όπου έχουμε άλλα πολλά προβλήματα και για τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος θα πρέπει τελικά να αυξήσουμε ε, ε, την ικανότητα ε, του Επιτρόπου Πότοσνικ και της δίκησής του, τις δυνατότητες του να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που είναι πραγματικά και τα έρχονται εδώ υπό μορφή αναφορών στην Επιτροπή μας. Και μιλάμε εδώ για παραβάσεις κανόνων. Και πάλι σας συγχαίρω, κυρία Διαμεσολαβητά, για την εργασία σας και πάλι Κάνω έκκληση στην ε, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και στον Επίτροπο Πότοσνικ. Είναι ε, ε, καιρός να δράσουν και όχι να έχουμε αξιολογήσει post-mortem, διότι αυτό το θέμα του περιβάλλοντος είναι post-mortem. Συνάδελφος Γιάρ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι καταλαβαίνω τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, ο συνάδελφος για μένα διατύπωσε σωστά το πρόβλημα. Όταν λαμβάνονται μεγάλα μέτρα για κάποιο τέτοιο για κάποιο τέτοιο έργο, τότε η Κομισιόν θεωρεί ότι τα κράτη-μέλη θα τηρήσουν τους νόμους. Χαίρομαι για αυτή την καλή πίστη, αλλά Έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές αυτήν εδώ την Επιτροπή ότι όντως πολλές φορές τα κράτη-μέλη δεν το κάνουν αυτό. Και πραγματικά το έχω πει πολλές φορές, χρειαζόμαστε έναν τρόπο να, που να μπορούμε να ελέγχουμε την ε, ορθότητα, την ομιμότητα, την συμμόρφωση, να μπορούμε να το αποδεικνύουμε αυτό. Και έχουμε πολλές αιτήσει παρόμοιες με, με αυτήν εδώ που μόλις αναλύσαμε. Και ναι, πρέπει να εκπληρωθούν οι διατάξεις και να δούμε και να διαβεβαιώσουμε ότι λειτουργούν, λειτουργεί η νομοθεσία. Εδώ οι πολίτε απευθύνθηκαν σε εσά, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, για αυτό το πρόβλημα στη Βιέννη. ο διάλογος ανάμεσα σε Κομισιόν και στον Ευρωπαδημοσιολαβητή ήταν καλός. Αλλά η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε να είναι κατά την ταπεινή μου άποψη. Εσείς ως διαμεσολαβητής ε, χτίσατε μια γέφυρα διαβουλεύσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την κρέμισε. Και πραγματικά ε, δεν, ε, πρέπει να δημιουργηθεί, να υπάρχει αυτή η γέφυρα επικοινωνία των πολιτών και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να, γίνονται, ε, πρέπει να παρουσιάζονται και οι δύο όψεις του νομίσματος και οι δύο πλευρές. δεν μπορούμε να σταματάμε, να διακόπτουμε το διάλογο έτσι ξαφνικά. Και είναι πολύ δύσκολο όταν πολύ, έρχεται σε πολύ δύσκολη θέση, καταλαβαίνω, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, όταν γίνεται κάτι τέτοιο, όταν διακόπτεται ξαφνικά ο διάλογος. Και αυτό δεν είναι καλό για κανέναν, ιδιαίτερα για εκείνους που έχουν επηρεαστεί από αυτό. Yeah, Σας ευχαριστώ για την τοποθέτησή σας περί σύγκρουσης συμφερόντων. Ε, δεν θέλω να κάνω αυστηρά σχόλια. Έχω διοριστεί ως εισηγήτρια για την εκθεσή σας. Νομίζω ότι στα μελλοντικά μας σχέδια θα πρέπει να προτείνουμε μια αναθεώρηση. Δηλαδή θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την ομοθεσία της μελέτης αντικτύπου. Και να σας πω, είναι πραγματικά ντροπιαστικό ότι λένε στους πολίτες ότι γίνονται κάποια πράγματα και τελικά δεν γίνονται. Αναφερθήκατε στο post-mortem εδώ. Είπατε ότι είναι μια εκτίμηση post-mortem και είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο και τελικά δεν γίνεται. και πραγματικά ε, οι πολίτες πιστεύουν ότι κάποια πράγματα λαμβάνουν χώρα, αλλά τελικά δεν γίνονται. Δεν είναι σοβαρό αυτό. Μας ε, ενδιαφέρουν αυτές οι πληροφορίες, θέλουμε να τις λαμβάνουμε από την Κομισιόν, αλλά εμένα δεν θέμα, ικανοποιήσω και τόσο πολύ να βγω και να πω αυτή την ιστορία, γιατί δεν είναι και τόσο πολύ καλή. Πάντως σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ σε εμά, ε, γιατί πολύ συχνά οι πολίτες μας πιστεύουν ότι τελικά δεν έχει κανένα νόημα να προσφύγουν γιατί τελικά οι αρχές κάνουν ό,τι θέλουν. Και πραγματικά προκαλείται μεγάλη απογοήτευση. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον τρόπο που αντιδρούν τα θεσμικά όργανα. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, δεν ζητά άλλο το λόγο. Επομένως θα ξαναδώσω το λόγο στον Δημεσολαβητή για να απαντήσει. I want you to know the Ombudsman does Κοιτάξτε, δεν έχω εξωγήινες δυνάμεις, να σας το πω αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της ε, Επιτροπής για τις αντιδράσεις τους και για την υποστήριξή τους. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να προσπαθήσω να απαντήσω ορισμένα σχόλια, να απαντήσω στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, γιατί παίρνω πάρα πολύ σοβαρά την προσπαθία σας να προσπαθήσετε να αποσαφηνίσετε το ζήτημα. Να σας πω δύο πράγματα δημοσίως. Όπως άκουσε ήδη και το όργανο αυτό, έχω πάρα πολύ καλές ε, σχέσεις με την Κομισιόν ε, στην πλειονότητα των υποθέσεων. Και έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις με την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Περιβάλλοντος. Ο κ. Φάνκερμπερκ ε, είναι πάρα πολύ καλός γενικός διευθυντής και έχει συνεργαστεί πάρα πολύ καλά με τον Ευρωπαϊκό Μεσολαβητή και προσπαθεί να υποφεληθεί από το δίκτυο των Ευρω... του Ευρωπαϊκού Συλλοβητή για να προσπαθήσει να επιλύσει ζητήματα που είναι σημαντικά για την Κομισιόν έτσι ώστε να μην ε, φτάσουν στη δική σας κλίμακα. Και γι' αυτό ακριβώς του διαθέτουμε το δίκτυο. Έτσι λοιπόν αυτό αποτελεί απόδειξη και της δικής μας ε, βούληση για συνεργασία. Λεχθέντος αυτού να σα πω τα εξή. Έχω τρία σχόλια σε σχέση με όσα είπατε. Το βασικό πρόβλημα που είχα ήταν ότι μόλις έλαβα τις διαβεβαιώσεις ότι θα προωθούνταν τα πράγματα, είδα το φάκελο και δεν υπήρχε καμία απόδειξη, εγγραφή που να προτείνει ότι τα υλοποίησατε λεφτά. Και πραγματικά αντιμετωπίζω πρόβλημα όταν εγώ πρέπει να έρθω και να αναφέρω εδώ σε αυτό το θεσμικό όργανο Υπήρξαν προφορικές κοινοποίησεις, δεν το αμφισβητώ, αλλά προφανώς και η δική μου δουλειά απαιτεί να βασίζομαι σε γραπτά κείμενα για να μπορώ να τα διαβιβάσω και στις άλλες πλευρές και δεν μπορούσα να διαβιβάσω στην άλλη πλευρά καμία διαβεβαίωση εφόσον δεν είχα γραπτές αποδείξεις. Από τη σκοπιά αυτή λοιπόν. <laughs> Κατανοώ το πόσο σας περιορίζει ο νόμος αλλά το θέμα δεν είναι μόνο ο νόμος, είναι και καλή διοίκηση. Και εγώ βρήκα ότι σε επίπεδο καλής διοίκησης, χρηστής διοίκησης, ήταν ελλειπής η απάντησή σας. Αυτό ήθελα να πω, δεν ήθελα να καταναλώσω πολύ χρόνο. Σίγουρα ο διαμεσολαβητής ποτέ δεν περίμενε, ούτε πρότεινε, ούτε ζήτησε η Κομισιό να προχωρήσει να, βάσει, να προσπαθήσει να κατεδαφίσει φυστάμενα κτίριο. Στη συστασή μου ποτέ δεν είπα κάτι τέτοιο. Απλώς αναφέρθηκα στο πώς θα διχειριστούμε μία καταγγελία, μία προσφυγή από πολίτες στο αυστριακό κράτος που είπαν ότι δεν μας δόθηκε δυνατότητα να έχουμε μία αναθεώρηση γιατί δεν το επιτρέπει το αυστριακό δίκαιο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και κατόπιν ανέμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να βρει μία λύση που να συνάδει με τη χρηστή διοίκηση και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι Κομισιόν και οι μα έχουν δείξει πόσο εφηβρητικές μπορούν να είναι όταν το επιθυμούν. Χωρί φυσικά να παραβιάζουν την νομοθεσία. Και εγώ θεώρησα ότι αυτή η συγκεκριμένη κατάσταση σε αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω να πιστεύω ότι πράγματι υπάρχει εδώ σύγκρουση συμφερόντων όταν ένα Υπουργείο της Δημοκρατίας της Αυστρίας είναι και αυτός που εκδίδει τις άδειε για τα κτίρια αυτά και το όργανο που εκδίδει τις άδειε, αλλά λέει και τίποτα δεν μπορεί να γίνει γι' αυτό. Νομίζω ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων λοιπόν εδώ. Και εγώ κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η απάντηση της Κομισιόν στο σημείο αυτό δεν ήταν αρκετά πιστική ότι οι προσφεύγοντες, οι καταγγέλλοντες είχαν κάνει λάθος. Αυτό ήθελα να πω. Τώρα δεν είναι πλέον στα χέρια μου το ζήτημα αυτό. Αυτό το θεσμικό όργανο θα αποφασίσει πώς θέλει να συνεχίσει, όμως εγώ ήθελα να το ξεκαθαρίσω αυτό το σημείο. Σας ευχαριστούμε και πάλι. θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε στην υπόθεση αυτή με τη δέουσα προσοχή και σοβαρότητα. Όπως σας είπα, οι πράσινοι θα αναλάβουν την έκθεση αυτή. Κύριε Διαμαντούρο, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ, σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία, συγχαρητήρια για το έργο σας και θα σας απελευθερώσω στο σημείο αυτό. Σας ευχαριστώ και εγώ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα. No, all right. ο, <laughs> ε, συνάδελφοι παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πάμε στο θέμα 18 για τα προβλήματα των, ε, των ευρωπαϊκών σχολείων θα μας μιλήσει η κυρία Αναγκόρη αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Αναγκόρα και είμαι πρόεδρος της Interparents και εκπροσωπούμε και συντονίζομαι τις ενώσεις γονέων για τα ευρωπαϊκά σχολεία και είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην ομάδα, στις ομάδες εργασίας. Συνοδεύομαι από μέλη της Επιτροπής Interparents, από τις Βρυξέλλες 1, Βρυξέλλες 2 και εκπρόσωπο που ασχολείται με τις ειδικέ εκπαιδευτικές ανάγκες του συστήματος και αν έχετε ερωτήσεις αργότερα ε, θα είμαστε διατεθειμένοι να απαντήσουμε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που έγινε πριν από ένα έτος όταν πολλοί γονείς, ε, μαθητές ε, και εκπαιδευτικοί διαδήλωσαν στις Βρυξέλλες, Λουξεμβούργος και σε πολλά άλλα μέρη για εναντίον των νέων μέτρων που εισήχθηκαν ούτως ώστε να γίνουν περικοπές ε, προϋπολογισμού και οικονομίας ε, στο σύστημα αυτό το εκπαιδευτικό. Το 2011 είχαμε μια περικοπή 7 εκατομμυρίων. Την επόμενο έτος ε, η Κομισιόν επέμενε να υπάρχει μηδενική αύξηση και ζήτησαν από το σχολείο να κάνουν εκτιμήσεις τα σχολεία ούτως ώστε να υπάρχει ε, μια ε, σταθερή ζήτηση. Αυτό είναι αντίθετο προς την ιδέα του balancing budget ε, της σύμβασης. Για να καλυφθεί το κενό έπρεπε να ληφθούν αποφάσεις για το πού θα βρεθούν, θα γίνουν οι οικονομίες και βρεθήκανε με την αναδιοργάνωση των μαθημάτων, την μείωση συντονισμού, την μείωση των ορών διδασκαλίας και επίσης των, των ε, στηριγμάτων ε, εκμάθησης ή ε, τα άτομα της κατηγορίας 3 δεν μπορούσαν να έχουν μαθήματα μητρικής γλώσσας εκεί όπου υπήρχαν. Αυτό ήταν ένας εξορθολογισμός και ξέρετε όλοι σήμερα τι σημαίνει αυτό και αυτό στην πραγματικότητα επηρέασε τα βασικούς τομείς εκπαίδευσης και εθίγησαν κυρίως τα μικρότερα τμήματα και οι μικρές γλώσσες και τα πιο ευάλωτα παιδιά που θέλουν επιπλέον βοήθεια και τις επιστήμες όπου δεν μπορούμε να έχουμε πολλά παιδιά σε ένα τμήμα. Στην, στο γαλλικό τμήμα δεν υπήρχαν αρκετοί μαθητές για την χημεία στα γαλλικά Γι' αυτό ε, το αγγλικό τμήμα έπρεπε να αναλάβει τη χημεία, ε, γιατί δεν υπήρχαν αρκετοί ε, ε, για τα προχωρημένα μαθηματικά, αρκετοί γαλλόφωνοι έπρεπε να πάνε στο γερμανόφωνο τμήμα. Αυτά, αυτές είναι οι προκλήσεις σήμερα, είναι ένα παράδειγμα, γιατί είναι δύσκολο να γίνουν οι οικονομίες. Οι προϋπολογισμοί των σχολείων δεν έχουν επιπλέον χρήματα, 84% καλύπτονται από μισθούς ε, των ε, εκπαιδευτικών και εκεί θα πρέπει να μειωθούν οι μισθοί για να γίνουν οι οικονομίες Έχουμε αυτό το έγγραφο 33 και διαμαρτυρήθηκαν οι γονείς και υπέγραψαν την αναφορά. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που πέρσι τον Ιούλιο, 12 Ιούλιο ακούσατε την αναφορά μας και για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που προκλήθηκε. Ήταν μια καμπή για τα ευρωπαϊκά σχολεία είδαμε ότι κατέρευσαν τα οικονομικά των σχολείων και η αντισταθμιστική ε, συνεισφορά δεν προβλέπεται πλέον ε, στην ε, σύμβαση και δεν είχαμε κανένα σεβασμό για την παιδαγωγική ακαιρεότητα του συστήματος, πράγμα που έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις πάνω στην εκπαίδευση. Δεν μπορεί κανείς να αφαιρεί, να προσθέτει και να αφαιρεί εκπαίδευση τόσο εύκολα. Θα πρέπει λοιπόν το σχέδιο αυτό να διαφυλαχθεί και ζητούμε να υπάρχει ένας έλεγχος εξωτερικός ανεξάρτητος σχετικά με το πρόγραμμα των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Για την ώρα η Επιτροπή που είναι υπεύθυνη για τα ευρωπαϊκά σχολεία είναι η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων ε, και βεβαίως ε, δεν ε, τίνει να λαμβάνει παιδαγωγικές αποφάσεις. Με ενδιαφέρον ακούσαμε τώρα τον διαμεσολαβητή. Θέλουμε λοιπόν έναν έλεγχο εξωτερικό, αυτόνομο, ανεξάρτητο το γεγονός που η Κομισιό απέτυχε να οργανώσει έναν τέτοιο έλεγχο ε, ε, αποτελεί ε, παράδειγμα κακοδιοίκησης όπως είπε ο διαμεσολαβητής και όλα αυτά αναφέρονται στα έγγραφα τα οποία έχετε ενώπιόν σας σήμερα. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θέλαμε να ζητήσουμε από την Επιτροπή Αναφορών. Θέλουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει έναν τέτοιο έλεγχο. Σχετικά τώρα με τον φετινό προϋπολογισμό βρισκόμαστε και πάλι σε μια κατάσταση όπου η Κομισιόν στη γνωμοδότησή της μπορούμε να έχουμε ένα εκατομμύριο λιγότερα από το balancing budget και παρά όλες τις προσπάθειες να κάνουν οικονομίες στα σχολεία βλέπουμε ότι είναι το τρίτο έτος περικοπών, το τρίτο έτος παγώματος Ε, μπορέσαμε να περικόψουμε 294 ε, που έχουμε ε, επιπλέον λοιπόν δαπάνες. 5,5 εκατομμύρια βρέθηκαν και περικόπηκαν και το προϋπολογισμό στο που θα έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι 173 εκατομμύρια αλλά θα θέλαμε να ζητήσουμε 100-180 εκατομμύρια που αρχικά είχαν θεωρηθεί ως αναγκαία για τη λειτουργία των σχολείων. Βεβαίως, η σημερινή συνειφορά έχει αυξηθεί σε πραγματικούς όρους, αλλά Αυτό οδήγησε σε άλλες μειώσεις στο σύστημα λόγω του γεγονότος τα κράτη-μέλη χρειάστηκε να μειώσουν τους μισθούς των ε, καθηγητών και ορισμένες αποσπάσεις. Έχουμε λοιπόν λιγότερα χρήματα που έρχονται από την Εθνική Οδό. Μπορώ να προβάλλω έναν πίνακα. Έχουμε λιγότερο ε, εισόδημα από τα δίδακτρα ε, διότι δεν υπάρχει αρκετός χώρος και επίσης η μισθή των εκπαιδευτικών ε, περιλαμβάνονται σε ένα νέο σχήμα που δεν έχει ακόμα τεθεί σε ισχύ. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα σχολεία δεν μπορούν να παρέχουν μια ποιοτική εκπαίδευση και δεν μπορούν να γίνουν βελτιώσεις σχετικά με τα προβλήματα συμφόρησης που υπάρχουν, τον υπερπληθυσμό των σχολείων. Ε, δεν μπορούν να υπάρξουν νέες εγκαταστάσεις. Βλέπουμε ότι έχουμε αύξηση του πληθυσμού, αύξηση δημογραφική, ε, αλλά συνεισφορά που μειώνεται. Ε, σε έναν πίνακα βλέπετε την κατανομή των οικονομικών έχει 59% η Επιτροπή, όχι η Επιτροπή, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν σταθερός 58-59% τα τελευταία χρόνια, ε, το μερίδιο των χωρών είναι 21% που είναι η εθνική μισθή τους οποίους ε, πληρώνουμε και αυτό μειώθηκε φέτος διότι όλο και ε, λιγότεροι ε, εκπαιδευτικοί είναι αποσπόμενοι και αυτό επιβαρύνει την συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ε, μειώσεις από τα δίδακτρα, μια μείωση 4% για την κατηγορία 2, 2% για την κατηγορία 3. Έχουμε λιγότερο εισόδημα που προέρχεται από τους γονείς, διότι δεν υπάρχει αρκετός χώρος ε, στα σχολεία για να δεχτούν τους μαθητές. Ε, θα ήθελα να τοποθετήσω σε ένα πλαίσιο, το πολιετές δημοσιονομικό ε, πλαίσιο. Περιλαμβάνονται τα σχολεία στην δίκηση που είναι 5,7 του συνολικού προϋπολογισμού και είναι λιγότερο του 2% τα σχολεία τα ευρωπαϊκά. Βλέπετε λοιπόν αυτό το μικρομερίδιο, μιλάμε για αυτό το πολύ μικρομερίδιο Γι' αυτό θα ήθελα ή δυνατόν να ζητήσουμε τον πραγματικό προϋπολογισμό 180 εκατομμυρίων που ανέφερα. Θα ήθελα να κλείσω αναφερόμενοι στην δικό σας ψήφισμα πέρσι, διότι πρέπει να, ε, να εξετάσουμε τα ευρωπαϊκά σχολεία και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπάθησε να το κάνουμε. Νομίζουμε ότι το γράμμα και το πνεύμα της σύμβασης υπονομεύονται, η συνεκτικότητα του συστήματος απελείται, οι περικοπές έχουν επιπτώσεις πάνω στα ουσιώδεις αρχές των ευρωπαϊκών σχολείων και θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα της διδασκαλίας και την ευζοία των μαθητών και επίσης απειλεί το μέλλον του συστήματος η ανισότητα διότι ε, δεν έχουν ορισμένες κατηγορίες μαθητών τις ίδιες παιδαγωγικές δυνατότητες. Αυτό εισάγει μια διάκριση που νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Θα θέλαμε ε, να επανέλθουμε στις 10 βασικές αρχές ε, των σχολείων του 53 που βλέπουμε στον ιστότοπο των ευρωπαϊκών σχολείων που ισχύουν σήμερα όταν, ε, όσο όταν άρχισαν τα ευρωπαϊκά σχολεία και γεννήθηκε η ιδέα της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης. Σύντομη περίληψη θα θέλαμε να αποκατασταθεί πραγματικός προϋπολογισμός με συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Θέλουμε να προσθεθούν τα 5,5 εκατομμύρια και θέλουμε το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο να ζητήσει αυτήν την εξωτερικό έλεγχο που είναι απαραίτητος για να διαβιλαχθεί η παιδαγωγική ποιότητα των σχολείων. Και τέλος, είμαστε εδώ και όλοι οι γονείς υπέγραψαν την αναφορά εδώ και ένα χρόνο διότι πιστεύουμε στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση και στην σημασία της και στο πνεύμα που διαβιβάζουν στα παιδιά μας τα ευρωπαϊκά σχολεία. Υπάρχουν επίσης δραστηριότητες πρόσθετες που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία και ζητούμε από τα κράτη-μέλη τα οποία είναι αποφασισμένα να επενδύσουν στην ε, παιδεία και στην ποιοτική εκπαίδευση και κινητικότητα να εφαρμόσουν, την αρχή αυτή στα ευρωπαϊκά σχολεία. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Σας ευχαριστώ για τις εξηγήσεις σας. Η Επιτροπή τώρα. Ο κύριος Μαρκουμπέρτο Μορούκα. Thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να ανακεφαλαιώσω, να σας πω ποια είναι η κατάσταση που οδήγησε στις αποφάσεις που συζητούμε εδώ σήμερα. Όλο αυτό το θέμα ξεκίνησε με την ψηφίση του προπολογισμού του 2011 η Δημοσιονομική Αρχή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφάσισαν το 2010 να κατανέμουν στα ευρωπαϊκά σχολεία 164 εκατομμύρια ευρώ ως συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί 171 εκατομμυρίων ευρώ που η Κομισιόν είχε ζητήσει στο προσχέδιο προπολογισμού. Σε σύγκριση με το 2010 η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωση, παρόλα αυτά αυξήθηκε κατά 6,5% σε σχέση με το μειωμένο νούμερο του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Είχαμε αύξηση 10, 10 εκατομμύρια σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ ο συνολικός δικαιωτικός προϋπολογισμός αυξήθηκε 2,9 Είχαμε λοιπόν διπλή αύξηση του διοικητικού προπολογισμού. Ο συνολικό προπολογισμό των ε, συστήματο των Ευρωπαϊκών Σχολείων αυξήθηκε 1,3%. Έτσι λοιπόν είναι πραγματικά δύσκολο να μιλήσουμε για περικοπές στον προπολογισμό. Το 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων έλαβε κάποια μέτρα για να βελτιστοποιήσει τη χρήση των πόρων που είχε στη διάθεσή του προσαρμόζοντας τους μισθούς ε, των ε, εκπαιδευτικών ε, και να υπενθυμίσω ότι οι μισθοί των εκπαιδευτικών έχουν ένα κανόνα παραλληλισμού με, το κανονισμό, με το μισθό των Ευρωπαίων υπαλλήλων. Ευτυχώ για τους δασκάλους η μεταρρύθμιση του 2004 που υιοθετήθηκε και εφαρμόστηκε για τους ε, υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ε, είχε ε, εφαρμοστεί για τους ευρωπαϊκούς εκπαιδευτικούς και βάσει της αρχής του παραλληλισμού τα ευρωπαϊκά σχολεία αποφάσισαν να εφαρμόσουν την ίδια μεταρρύθμιση προκειμένου τα δύο συστήματα να είναι παράλληλα. Και αυξάνοντας το κατόφλι σε ό,τι αφορά τον πληθυσμό στις τάξεις. Αυτό προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις ε, και στα σχολεία του Λουξεμβούργου 1 και Βρυξέλλες 1 ε, υπήρξε ο φόβος ε, ότι η αύξηση του αριθμού των μαθητών ε, θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα των μαθημάτων. Το 2012 τώρα μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα μέτρα που ελήφθησαν το 2011 για τη μείωση των δαπανών των ευρωπαϊκών σχολείων ήταν επιτυχή. Τα ευρωπαϊκά σχολεία δεν, έπρεπε να, δεν χρειάστηκε να ζητήσω συμπληρωματικό προπολογισμό και τα μέτρα δεν ε, μείωσαν την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται στα σχολεία. Σε ό,τι αφορά τώρα τα αιτήματα που παρουσιάστηκαν σήμερα από την ε, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων, υπήρξε μια ανησυχία σε σχέση με έναν έλεγχο και η Κομισιόν ε, ε, συμφωνεί πλήρως ε, με το Σύλλογο Γονέων. Έγινε ήδη ένας έλεγχος από το σύστημα PISA του ΟΣΑ για το σχολείο του Ξεμβούργου. Τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ θετικά και είμαστε σε επαφή με τον ΩΣΑ για να κάνουμε έναν έλεγχο για όλο το σύστημα των ευρωπαϊκών σχολείων. Έτσι λοιπόν, ανυπομονούμε να υλοποιηθεί ο έλεγχος αυτός. Ε, για το σχολείο του Λουξεμβούργου ήταν πάρα πολύ καλά τα αποτελέσματα σε σχέση με το μέσο όρο των υπόλοιπων σχολείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τώρα τον προπολογισμό το φετινό, που παρουσιάστηκε βάσει μιας αναφορά του 2011. Υπάρχει όμω και ένα νέο θέμα που αφορά το φετινό προπολογισμό. Να τονίσω ότι η Κομισιόν ζήτησε αύξηση 5,1% του προϋπολογισμού σε σχέση με πέρσι και στη σύγκριση αυτή βλέπουμε ότι ο διοικητικός προϋπολογισμός έχει απλώς παγώσει Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση όπου έχουμε διοικητικό προπολογισμό 0% για τις διοικητικές δαπάνες και τα σχολεία έχουν 5% αύξηση. Νομίζω ότι υπάρχει μια μικρή παρανόηση για το θέμα της ε, εξισορρόπησης των εισφορών. Το σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων είναι ένα σύστημα που βασίζεται και στις εισφορές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως και έτσι ψηφίστηκε από το Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο που εκπροσωπούνται όλα τα κράτη-μέλη. Και πρέπει να τονίσω ότι ο τελικός προϋπολογισμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων εθετείται μόνο όταν η Δημοσιονομική Αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει οθετήσει το δικό της προϋπολογισμό όσο η Δημοσιονομική Αρχή δεν έχει αποφασίσει επί της συνεισφοράς, τα ευρωπαϊκά σχολεία δεν έχουν υιοθετημένο ένα τελικό προϋπολογισμό. Δηλαδή, υπάρχει εξισορρόπηση της συνεισφοράς Ε, υπάρχει εξισορρόπηση για το τμήμα που δεν δίνεται από τα κρατη και για τις άλλες πηγές εισοδήματος για τα ευρωπαϊκά σχολεία. Όμως η Δημοσιονομική Αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, έχουν την πλήρη εξουσία στο θέμα αυτό. Άλλο ένα θέμα τέθηκε, υπερπληθυσμός της τάξης και της μη απόσπασης των εκπαιδευτικών. Να ξεκινήσω από το δεύτερο, της μη απόσπασης. πραγματικά αυτό όθησε το σύστημα στα όρια του, γιατί είναι απαραίτητη η εκπαιδευτική για δύο λόγους. Φυσικά για να διδάξουν σε ένα σχολείο, αλλά και η αποσπασμένη εκπαιδευτική είναι απαραίτητη γιατί επιτρέπουν μια συνεχή διαβίβαση γνώσης από τα εθνικά συστήματα στα ευρωπαϊκά σχολεία, στο σύστημα των ευρωπαϊκών σχολείων. Έτσι λοιπόν η απόφαση ορισμένων κρατών μελών να μειώσουν τον αριθμό των ασφασθέντων είναι πολύ επικίνδυνη και είναι και πάρα στα πολύ επικίνδυνη για τους σπόρους του σχολείου. Γιατί αν δεν αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, τότε το ευρωπαϊκό σύστημα αναγκάζεται, θα αναγκαστεί να προσλάβει τοπικά εκπαιδευτικούς, εκεί δηλαδή όπου είναι εγκαταστημένα τα ευρωπαϊκά σχολεία, γενικά καλή είναι αυτή η εκπαιδευτική, αλλά η ποιότητα των εκπαιδευτικών που προέρχονται από τα κράτη-μέλη, καθώς έχουν επιλεχθεί ειδικά και έχουν υποστεί και ειδική κατάρτιση, είναι άλλης αξίας. Έτσι λοιπόν η Κομισιόν βασίζεται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην ε, αρμοδιότητά του να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να συνεχίζουν να αποσπούν πολλούς εκπαιδευτικούς στο σύστημα των ευρωπαϊκών σχολείων. Τουλάχιστον αυτούς που θα πρέπει να στείλουν ε, βάση του αναλογικού κανόνα, όπως τον αποκαλούμε. Δηλαδή να έχουμε ανάλογο αριθμό δασκάλων με τον αριθμό των μαθητών. Κατόπιν, έχουμε το θέμα του υπερπληθυσμού. το ζήτημα. Σε πολλά σχολεία, κυρίως ε, στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο έχουμε υπερπληθυσμό και ακόμη και αν θα βελτιωθεί κάπως η κατάσταση φέτος, καθώς ε, ε, θα ανοίξουν νέα σχολεία, δεν θα επιληθεί ε, το Συμβούλιο ζήτησε και για πέμπτο σχολείο στις Βρυξέλλες, αλλά οι διαπραγματεύσεις ε, εξακολουθούν να είναι σε εξέλιξη με τα κράτη-μέλη και με το Βέλγιο και δυστυχώς το Βέλγιο ακόμη δεν μας έχει δώσει μια τοποθεσία για το πέμπτο σχολείο. Αυτό πρέπει να λάβει χώρα σύντομα προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για τους μαθητές μας. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, κάποιος συνάδελφος θα ήθελε να παρέμβει. Ναι κύριε Γιάρη. Ευχαριστώ πολύ. Από ό,τι βλέπετε και αυτή η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολήθηκε με αυτό το πρόβλημα, ιδιαίτερα η επιτροπή που χαρακτήρισε και αυτή την αναφορά ως επίγουσα. Και έγινε έτοιμα για ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχουμε ένα πρόβλημα. Μπορούμε να δούμε πολιτικά το θέμα. Και πολιτικά το θέμα είναι ξεκάθαρο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μιλήσει σαφέστατα για το ζήτημα αυτό, για... έχει ζητήσει τη χρηματοδότηση τους και το μοντέλο και η ιδέα θεωρείται εξαιρετικό, θεωρείται κατάλληλο. Και βλέπω τώρα ότι κάνουμε κύκλους γύρω από το ζήτημα αυτό. Είπα είναι μια ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργηθούν αυτά τα ευρωπαϊκά σχολεία. Έχει χρηματοδοτηθεί από τον ε, προϋπολογισμό, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. Και εδώ συζητούμε την ποιότητα και, ε, και το πρόβλημα που έχουμε με την ποιότητα σε αυτά τα ευρωπαϊκά σχολεία. Το Κοινοβούλιο έχει συμφωνήσει, όχι 100%, 200% για αυτά τα ευρωπαϊκά σχολεία, για την αύξηση της ποιότητας. Εδώ Πιστεύω πως είναι αναγκαία μια εξωτερική, ανεξάρτητη, ένας ανεξάρτητος εξωτερικός εμπειρογνώμονας, ο οποίος θα κάνει εκτενής ανάλυση αυτών των σχολείων, για να δούμε και φυσικά η Κομισιόν έχει πει ότι υπάρχει ε, υπερπληρότητα των σχολείων αυτών, έχει διαπιστωθεί αυτό, αλλά πρέπει να εξετάσουμε τα θεμέλια, να δούμε πού βρισκόμαστε, τι χρειαζόμαστε, τι μας λείπει. Πρέπει λοιπόν να γίνει αυτή η ανάλυση εμπειρογνωμόνων, να δοθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμού, να, η οποία θα εξάγει στη συνέχεια συμπεράσματα και στην τελευταία συνεδρίαση ανέφερα ότι θα έπρεπε να ενημερώσουμε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να τους ενημερώσουμε και για τις υποχρεώσεις τους. Δημιουργήθηκαν λοιπόν αυτά τα ευρωπαϊκά σχολεία, αλλά απομακρύνονται από τις υποχρεώσεις τους ανά ένα τα μελη Και πραγματικά, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύω ότι είναι υποχρεώσή μας να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Γιάρ. Ο κύριος Έφνες ζήτησε το λόγο. Αγαπητέ Πίτερ, μπορώ να σας να συμμετέχω κι εγώ. Δεν μπορώ να κάνω ταχυδακτουλουργικά κόλπα, αλλά είναι σίγουρο ότι τα ευρωπαϊκά σχολεία και αυτό είναι από την εμπειρία μου με ανθρώπους που στέλνουν τα παιδιά τους εκεί, που κάνουν εξαιρετικό μεν έργο, αλλά πραγματικά έχουν πρόβλημα, είναι υπερπλήρη. Και επίσης είναι, σίγου, είναι γεγονός ότι τα προβλήματα και οι δεσμεύσει του προϋπολογισμού που αναφέρθηκαν έχουν φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να προχωρήσουμε άλλο. Δεν μπορούμε εμείς όμως να λάβουμε αποφάσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό τους. Ε, σωστό και συνετό είναι, όπως πρότεινε και ο Πίτερ στο παρελθόν, να μεταφερθεί το ζήτημα αυτό στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Με την παράκληση να το κοιτάξουν, διότι εκείνοι έχουν, ε, μπορούν να επηρεάσουν τον προϋπολογισμό. Μπορούν να κάνουν κάτι, μπορούν να κάνουν αξιολογήσεις και να δουν τι, μπορούν, τι μπορεί να αλλάξει, τι μπορεί να βελτιωθεί. Ε, εγώ δεν μπορώ να σας πω κάτι τώρα έτσι στα γρήγορα όμως είμαι σίγουρος ότι η Επιτροπή αυτή είναι πιο αρμόδια και μπορεί να δώσει λύσεις. Ε, ε, και στους δύο και στην πρόεδρο των Into και στην, στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Ε, για το 2012 λέτε ότι η Δημοσιονομική Αρχή δεν έχει ακόμα αποφανθεί για τα ποσά που ετήθηκε η Επιτροπή και ένα από τα οποία έχει σχέση με τα σχολεία. Ε, ε, αυτό το γνωρίζετε και οι δυο. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση μέσα στον Αύγουστο να γνωρίζουμε τι ποσό μπορεί να, πάρει, να πάρουν τα ευρωπαϊκά σχολεία. Uh, Αν σας κατάλαβα καλά, συζητούμε τα ποσά για το 2013 που θα συζητηθούν τώρα. Η Κομισιόν παρουσίασε το νούμερο 173,8 εκατομμύρια και ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ως δημοσιονομικές αρχές θα εγκρίνουν αυτό το νούμερο. Είναι το νούμερο που ομόφωνα υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο των Κρατών Μελών. And, uh, Οι interparents ε, θα ήθελαν να ζητηθούν 180 εκατομμύρια που αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δημοσιονομικές ανάγκες των σχολείων παρά αυτό που υιοθετήθηκε. Πάρα πολύ. Ε, εκτιμώ η πρόταση του κυρίου Γιάρ. Α. Ας συνοψίσω ξανά την πρόταση. Τα σχολεία καταστρο... καταρτούν το σχέδιό τους για όλων των χρόνων, για το... το στην ημερολογιακή χρονιά, όχι την ακαδημαϊκή, τη σχολική χρονιά. Και αυτό δεν, δεν, ε, είναι, δεν συνάδει με την, με την κατάρτιση του προϋπολογισμού, η οποία γίνεται σε ημερολογιακά ετήσια βάση. Μιλάμε τώρα για το Σεπτέμβριο, για το νέο σχολικό έτος, και ήδη έχουμε φτάσει στο 2013, δηλαδή υπάρχει μία διαφορά. Συνοψίζοντας, η αίτηση αυτή προτείνω να μεταφερθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμού και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού με την παράκληση να ασχοληθούν μαζί της επιγόντως και να γίνει μια αντικειμενική εξέταση εμπειρογνωμόνων, να γίνουν εκθέσεις εμπειρογνωμόνων για να λυθεί αυτός αυτό το κουβάρι που έχουμε εδώ μπροστά μας. Για να μας δοθούν απαντήσεις. Και επίσης, όπως είπα, πολιτικά υπάρχει η συμφωνία. Υπάρχει η, συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ευρωπαϊκά, ευρωπαϊκά σχολεία. Όσον αφορά τώρα τα οικονομικά ζητήματα, το ζήτημα της χρηματοδότησης, δεν είμαστε εμείς η αρμόδια επιτροπή. Πρέπει να το φέρουμε το ζήτημα στο κατάλληλο επίπεδο, στους αρμόδιους. Διότι εκείνοι μπορούν να μας ξεκαθαρίσουν τις ε, ασάφειες που εμείς δεν μπορούμε να λύσουμε. Να δούμε τι γίνεται με τον, στον περιπολογισμό του 2013. Αυτή θα ήταν η πρότασή μου, την αφήνω ανοιχτή για τα σχόλια και για συζήτηση και πραγματικά ε, επιθυμώ να παραμείνουμε ανοιχτοί και να ε, έχουμε επικοινωνία αλλά όπως είπα να επιστήσουμε την προσοχή στο επίγον του ζητήματος στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Διότι αυτό αφορά όχι μόνο τους μαθητές αλλά και τους εργαζόμενους στα σχολεία αυτά. Ευχαριστώ. Δεν υποστηρίζω μόνο τις προτάσεις ε, των κυρίων Γιάρ και Χέφνερ, αλλά θα ήθελα να προσπαθήσω να εμπλέξω και την Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, γιατί και αυτή η Επιτροπή έχει λόγο για το ζήτημα αυτό και κατόπιν να σκεφτούμε αν εμείς ως Ευρώπη δεν είμαστε σε θέση να καλύψουμε τις ανάγκες των ευρωπαϊκών σχολείων πώς θα φανταστούμε ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για να αυξήσουμε περαιτέρω την προβολή και την εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό Κοδόμημα και πώς ε, θα προετοιμάσουμε το μέλλον. Όταν ε, μιλάμε ότι εργαζόμαστε για του κοινού ευρωπαϊκού στόχου αυτό είναι και ο τρόπο να προετοιμαστούμε για το ευρωπαϊκό μα μέλλον, ε, τώρα που είμαστε μεσούσες της κρίσης. Δεν μπορούμε να μεταχειριζόμαστε τα ευρωπαϊκά σχολεία με την ίδια συνταγή λιτότητα, λιτότητα, λιτότητα. Γιατί η λιτότητα είναι καλή, αλλά δεν αρκεί. Πρέπει να προσθέσουμε και κάτι στη λιτότητα. Και για τους μαθητές αυτό είναι θεμελιώδες. Νομίζω ότι όλοι τα ίδια πιστεύουμε εδώ, είμαστε ενωμένοι και μπορούμε να υποστηρίξουμε να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, να σταλεί στην Επιτροπή Προπολογισμού και στην Επιτροπή Πολιτισμού και να δούμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε. Ίσως θα μπορούσαμε να τη διαβάσουμε και στη διάσκεψη των Προέδρων, γιατί είναι επίγον το μήνυμα αυτό, γιατί ε, ουσιαστικά δεν μπορούμε να προβλέψουμε το 2013, τον προπολογισμό του 2013, χωρί να δίνονται τα απαραίτητα κονδύλια ε, που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό χωρί να έχουμε μια προβλεψιμότητα και για το μέλλον. Και η προβλεψιμότητα τι σημαίνει. Πρέπει να έχουμε έναν αξιοπρεπή προπολογισμό. Ανακεφαλαιώνω. Κρατούμε την ε, αναφορά ανοιχτή ε, με βάση τις προτάσεις ε, του κ. Γιάρ και τη δική σας κ. Μποστινάρου θα στείλουμε ε, το θέμα στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και Ελέγχου Προϋπολογισμού και βεβαίως και στην Επιτροπή ΚΑΛΤ στην οποία υπάγεται το θέμα στην ουσία του. Εγώ θα ήμουν ευτυχής ο θεσμός να υιοθετηθεί από όλα τα κράτη-μέλη ως ένα πρότυπο σωστής εκπαίδευσης που μπορεί να λειτουργήσει ως μοντέλο. Λοιπόν, αυτή ήταν παρέτηση και προτείνω επίσης να τα στείλουμε και στο Council και στο, και στο Συμβούλιο γιατί τους αφορά όλους προς αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, όχι μόνο στις τρεις επιτροπές αλλά και στο Συμβούλιο. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να πάνε καλύτερα του χρόνου. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Προχωρούμε στο επόμενο θέμα. Κάνουμε μια μικρή αλλαγή στην ε, ε ημερήσια διάταξη. Πάμε στην petition ε, αριθμός 20 ε, από τον κύριο Κέμπεν εκ μέρους ε, που αντιπροσωπεύει... Ε, είναι παρόν ο κύριος Μπέρναρ Κέμπεν. Ja ich bin anwesend. Μάλιστα είμαι εδώ. μπορεί να κινήσετε κιόλας. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί Ευρωβουλευτές, Αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω για τους εκ των υπολείπων επιχειρήσεων. Ε, θα σας μιλήσω ιδιαίτερα για την φίρμα BPM και θέλω να σας στην προσοχή σας σε δύο πράγματα. Η εταιρεία αυτή έχει την έδρα της στη Βιέννη και είναι λοιπόν υποχρεωμένη να εγγραφεί στο ε, εμπορικό επιμελητήριο της Αυστρίας. Ανοίγοντα ένα παράρτημα στο Βερολίνο, με προς έκπληξή μας διαπιστώσαμε ότι η Γερμανία δεν εφαρμόζει την οδηγία για τις παροχές υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει τη διπλή εγγραφή σε επιμελητήρια. Έτσι λοιπόν εμείς αναγκαστήκαμε να εγγραφούμε και στο γερμανικό ε, βιομηχανικό και εμπορικό επιμελητήριο. Εγώ Προσωπικά από το 2004 είμαι μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου. Όταν επανεκλέχθηκα το 2009 έπρεπε η δική μου εκλογική ομάδα να έχει 167 ψήφους για να λάβει θέση σε αυτήν την συνέλευση των επιμελητηρίων. Δίπλα μου είχα άλλους συναδέλφους από άλλες εκλογικές ομάδες οι οποίοι χρειαζόντουσαν μόνο 21 και 25 ψήφους για να λάβουν έδρα. και πώς, μπορούν να δια, να, ε, πώς μπορούμε να διατηρήσουμε δημοκρατικά, ε, δημοκρατικά πρότυπα, πώς, πώς υπάρχει δημοκρατία σε αυτό. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά μου προκαλεί έκπληξη και σοκ. Ευχαριστώ. Να μας μιλήσουν από την Επιτροπή ο κύριος Δημητριάδη. Α, παρακαλώ. Αγαπητοί Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι ο κύριος Κέμπεν, ο συνάδελφος που μίλησε ήταν ο κύριος Μπέτιγχάους. Εγώ είμαι καθηγητής στο Πανεπιστημίο της Κολονίας. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που μου δώσατε την δυνατότητα εδώ να παρουσιάσω την αναφορά μας. Θα είμαι, προσπαθήσω να είμαι σύντομος και να αναφερθώ σε τέσσερα σημεία. Καταρχάς στην δομή και τις αρμοδιότητες του Γερμανικού Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου. Στη Γερμανία υπάρχουν χωρισμένα σε περιφερειακούς τομείς περίπου 80, συνολικά μάλλον 80 βιομηχανικά και εμπορικά επιμελητήρια. Και κάθε ελεύθερος επαγγελματίας, είτε το θέλει είτε όχι, είναι υποχρεωμένος με νόμο να είναι μέλος με υποχρέωση εισφορών στο επιμελητήριο της περιφέρειάς του. Κύριο έργο, κύρια αρμοδιότητα του μελητηρίου αυτού είναι και αυτό είναι ε, απόσπασμα από τον νόμο να αντιπροσωπεύει το συνολικό συμφέρον των μελών της περιφέρειάς του. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε με δημόσια διαμόρφωση απόψεων με, ε, που γίνεται από οργανισμούς δημοσίου δικαίου και μπορούμε να πούμε δηλαδή με λόμπι άσκησης πίεσης, μέσω λόμπι άσκησης πίεσης σύμφωνα με τον νόμο δεν είναι αρμοδιότητα των βιομηχανικών και εμπορικών επιμελητηρίων να δίνουν άδειε εξάσκηση επαγγέλματο και να λαμβάνουν αποφάσει σχετικά με αυτέ, να, να έχουν πειθαρχικέ αρμοδιότητε ή να ε, παρακολουθούν την τήρηση των επαγγελματικών προτύπων. Αυτό κάνει τη διαφορά ανάμεσα στο βιομηχανικό και εμπορικό επιμελητήριο και στα τεχνικά επιμελητήρια ή τα... τους ιατρικούς συλλόγους, τους δικηγορικούς συλλόγους, τους συλλόγους των φαρμακοποιών ή το επιμελητήριο για παράδειγμα των αρχιτεκτόνων. Έπειτα, δεύτερο σημείο, σχετικά με την μη δημοκρατική εσωτερική οργάνωση των βιομηχανικών και εμπορικών επιμελητηρίων. Οι ετώντες περιορισμένοι, αισθάνονται περιορισμένοι για την ακατάπαυστη δημόσια θέση των εμπορικών και ε, βιομηχανικών επιμελητηρίων σε όλα τα ζητήματα, σε όλα και περισσότερα ζητήματα. Για παράδειγμα, για την ενεργειακή πολιτική, για την οικονομική κρίση, για, ε, για διάφορα άλλα θέματα. Και οι ετώντε δεν έχουν καμία ευκαιρία, καμία δυνατότητα να παρουσιάσουν τι δικέ του θέσει, να προσπαθήσουν να ασκήσουν επιρροή στην διαμόρφωση βούληση των γενικών συνελεύσεων των επιμελητηρίων αυτών, διότι σύμφωνα με το ισχύον δικαίωμα εκλογής, την περισσότερη επιρροή στις γενικές συνελεύσεις των επιμελητηρίων τις έχουν εκείνοι που, οι επιχειρήσει που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα κέρδη. Για να σα δώσω ένα παράδειγμα. Η Γενική Συνέλευση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της πόλης Braunschweig απαρτίζεται από 80 αντιπροσώπους. Ο ετών στο, στην περίπτωση 4, ένα σύμβουλος επιχειρήσεων έχει δικαίωμα ψήφου μόνο στην ομάδα των παρόχων υπηρεσιών και αυτή η ομάδα μπορεί να στείλει 5 αντιπροσώπους στην Γενική Συνέλευση του Μελητηρίου. Ένας βιοτέχνης έχει ταυτόχρονα 17 αντιπροσώπους και ένας βιομήχανος 26 αντιπροσώπους στην ίδια Γενική Συνέλευση. Και αυτό, κατά την άποψη των ε, ετώμενων, είναι αναχρονιστικό και βαθιά μη δημοκρατικό δικαίωμα ψηφοφορίας. Τρίτο σημείο για την ελευθερία εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών. Η υποχρεωτική συμμετοχή πιστεύουμε ότι παραβιάζει την, ε, την ελευθερία εγκατάστασης, την ελευθερία παροχής υπηρεσιών και την οδηγία παροχής υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ακόμα δεν έχει λάβει αποφάσεις για αυτό. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μέχρι τώρα έχει λάβει αποφάσεις για την υποχρεωτική ε, εγγραφή στα αυτορυθμιζόμενα επιμελητήρια, δηλαδή στα βιοτεχνικά επιμελητήρια, στους δικηγορικούς συλλόγους και στους συλλόγους εκτινιάτρων, όχι όμως ακόμα για την υποχρεωτική εγγραφή στα βιομηχανικά και εμπορικά επιμελητήρια. Στα αυτορυθμιζόμενα επιμελητήρια, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είδε δικαιολόγηση ε, για την, παρέμβαση στην ε, ελευθερία εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών στα συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα καθήκοντα αυτών των επιμελητηρίων. Επιμελητήρια τα οποία υπηρετούν τους πελάτες, τους ε, ασθενείς ή τους καταναλωτές και αυτή η δικαιολόγηση λόγω μη συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων που έχουν διάφορα λόμπι δεν μπορεί να μεταφερθεί στα ε, βιομηχανικά και εμπορικά επιμελητήρια. Επίσης, είναι προφανές προφανής η παράβαση στην, ε, εντολή, στην οδηγία παροχής υπηρεσιών, η οποία ρητά απαγορεύει διπλή εγγραφή σε δύο κράτη-μέλη. Και αυτή η διπλή εγγραφή όμως είναι, ήταν γεγονός στην περίπτωση του αυστριακού αναφέροντος. Είναι μέλος δηλαδή του ε, βιομηχανικού επιμελητηρίου της Αυστρίας και ενός στη Γερμανία. Τέταρτο σημείο είναι μια σύντομη επισκόπηση της κατάστασης ε, στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια τέτοια υποχρεωτική εγγραφή σε επιμελητήριο όπως στην Γερμανία υπάρχει μόνο σε έξι κράτη-μέλη. Στην Γαλλία, στην Ιταλία, στις κάτω χώρες, στην Αυστρία, την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο. Ωστόσο, οι αρμοδιότητες των επιμελητηρίων αυτών διαφέρουν πάρα πολύ από εκείνος του γερμανικού επιμελητηρίου. Γι' αυτό δεν μπορούμε εμείς να πούμε εάν αυτή η υποχρέωση εγγραφή σε αυτά τα έξι κράτη-μέλη είναι... Ε, διαπράττει κάποια παράβαση ή έχει νομιμότητα. Μπορούμε να πούμε όμως, να μιλήσουμε για την κατάσταση στην Γερμανία και στην Αυστρία. Η Ισπανία μόλις ε, πριν από λίγο κατάργησε την υποχρεωτική εγγραφή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συστήνει την κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής και στη Γερμανία διότι παρακολύει κατά την άποψή τους την ε, οικονομική ανάπτυξη. Και τέλος κυρίες και κύριοι θα εκτιμούσα πάρα πολύ εάν η Επιτροπή Αναφορών ζητούσε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία ουσιαστική και επί της ουσίας γνωμοδότηση, καθώς επίσης και να ζητήσει από την Επιτροπή, την Νομική Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου να αναμειχθεί. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Τώρα ο κύριος Δημητριάδης, παρακαλώ. Thank you, Chair. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι το 2010 και 2011 λάβαμε πέντε προσφυγές ε, και ίσο αριθμό αναφορών ε, σχετικά με την υποχρεωτική εγγραφή ε, στα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια Αυστρίας και Γερμανίας. Είχαμε τέτοιες προσφυγές μόνο σχετικά με τη Γερμανία και την Αυστρία, όχι σχετικά με άλλες χώρες. Θα πρέπει ότι η αναφορά έγινε το 2010 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έλαβε ο αναφέρον μία απάντηση εξηγώντας γιατί η Επιτροπή δεν σκοπεύει να λάβει κανένα μέτρο σχετικά με την προσφυγή του. Και τώρα έχει ε, αναφερθεί ε, στην Επιτροπή Αναφορών όλες οι προσφυγές έκλεισαν, όλες οι αναφορές έκλεισαν, η προηγούμενη έκλεισε χωρίς ούτε καν συζήτηση. Τώρα, σχετικά με την ουσία, με την ουσία της αναφοράς και της προσφυγής θα πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, την ομολογία του δικαστηρίου δεν είναι υπέρ της αναφοράς. Η υποχρεωτική εγγραφή στα εμπορικά επιμελητήρια ε, δεν συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο που εγγυάται την ελευθερία της εγκατάστασης. Το δικαστήριο ήταν σαφές ότι σε περίπτωση ελεύθερης παροχής υπηρεσιών όταν μια επιχείρηση είναι κατεστημένη σε ένα κράτος μέλος και παρέχει υπηρεσία σε άλλο κράτος μέλος τότε η υποχρεωτική εγγραφή στο εμπορικό επιμελητήριο είναι τελείως ασυμβαστή με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Όμως, σε περίπτωση ελευθερίας εγκατάστασης, ο περιορισμός μπορεί να αιτιολογείται και, επομένω μπορεί να είναι συμμετό με το άρθρο 49. Δεν είναι μόνο όταν το εμπορικό επιμελητήριο ή ο ιατρικός σύλλογος έχει απλώς αρμοδιότητες για το θέμα της ηθικής ε, των μελών. Αυτή είναι μία από τις περιπτώσεις, αλλά έχουμε και την περίπτωση Κώστεν, όπου το δικαστήριο είπε ότι η υποχρεωτική εγγραφή ε, σε ένα επιμελητήριο παρόμοιο με το περιοικολογικό επιμελητήριο και η ε, πληρωμή της εγγραφής θα μπορούσε να αιτιολογηθεί στην περίπτωση του κράτους μόνης υποδοχής. Έτσι λοιπόν η νομολογία του δικαστηρίου δεν είναι ευνοϊκή στην αναφορά. Έτσι λοιπόν η Κομισιόν δεν μπορεί να αναλάβει περαιτέρω δράση για το θέμα αυτό. Πρέπει να δούμε ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Η υποχρεωτική εγγραφή στα εμπορικά επιμελητήρια είναι περιορισμός, μπορεί να είναι κάποιο μέλο και να μην κάνει τίποτα. Ποιο είναι ο πραγματικό περιορισμός. Ο πραγματικό περιορισμός είναι η πληρωμή τελών, η καταβολή τελών. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα των αναφερόντων. Γιατί στη Γερμανία και στην Αυστρία τα τέλη είναι αρκετά υψηλά. Κατανοούμε τους αναφέροντες ότι πρέπει να πληρώσουν πολλά χρήματα για κάτι που δεν θέλουν ή για υπηρεσίες που δεν θέλουν πραγματικά να λαμβάνουν. Είχαμε μια καταγγελία, μια προσφυγή ε, από έναν Γερμανό αυτοαποσχολούμενο που είπε ότι πρέπει να πληρώνω πάνω από 1000 ευρώ στο επιμενητήριο Τον βιοτεχνών. Έτσι λοιπόν πρέπει τουλάχιστον να εργάζομαι μία εβδομάδα για να πληρώνω αυτά τα χρήματα, ενώ ο Σλοβάκο συνάδελφο έρχεται εδώ για να παρέχει υπηρεσία στη Γερμανία και δεν πληρώνει τίποτα. Δεν είμαι ανταγωνιστικό λοιπόν εγώ. Και είχαμε και μία προσφυγή από μεγάλη αυστριακή εταιρεία με 60.000 εργαζομένους που είπε ότι πρέπει να πληρώσω 3,5 εκατομμύρια ευρώ ως τέλος εγγραφή. Είναι κατανοητό. Ότι φυσικά δεν θέλουν οι άνθρωποι να πληρώνουν ένα ποσό χρημάτων για κάτι. Για υπηρεσίες ή για οτιδήποτε δεν θέλουν να λαμβάνουν. Είναι λογικό ότι μεταξύ των εκατομμυρίων των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων στην Γερμανία είναι κάποιοι που δεν θέλουν να λαμβάνουν τις υπηρεσίες ε, του εμπορικού επιμελητηρίου. Προσφέρονται πάρα πολλές υπηρεσίες, νομική, αρρωγή ε, και άλλου είδους υπηρεσίες, κατάρτιση. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό κάτι τέτοιο, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα για την Κομισιόν και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα εθνικό πρόβλημα για τη Γερμανία και για την Αυστρία. Και υπάρχουν εθνικές κυβερνήσεις που υποθέτω ότι είναι έτοιμες να συζητήσουν το πρόβλημα και να βρουν μια λύση, αν είναι αρκετά υψηλά τα τέλη. Έτσι λοιπόν δεν είναι πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, νομίζω ότι είναι πρόβλημα σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή, οι αναφέροντε θα πρέπει να συζητήσουν το θέμα αυτό με τι αντίστοιχε εθνικέ κυβερνήσει και να προσπαθήσουν να εξεύρουν λύση. Στο πολιτικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιούνται. Σε ό,τι αφορά ορισμένε από τι παρατηρήσει. Ότι η λειτουργία των επιμελητηρίων δεν είναι δημοκρατική. Θα μπορούσε να υποθεί κάτι τέτοιο για τι δημοκρατίε μα. Ξέρετε, υπάρχουν ε, κάποιοι, το σχάρι, που εκπροσωπούν ε, λιγότερο από το 3% του πληθυσμού. Αυτά είναι προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει περιορισμό στην ελευθερία εγκατάσταση των εταιριών. Και φυσικά είναι και σημαντικό το ότι δεν έχουμε λάβει καμία προσφυγή, καμία καταγγελία από επαγγελματίε ή από εταιρείε που να έχουν εγκατασταθεί σε άλλο κράτο μέλο πέραν τη Αυστρία και τη Γερμανία ε, που δεν θέλουν να πάνε εκεί και να παραπονεθούν, να καταγγείλουν ότι περιορίζεται το δικαίωμα της εγκαταστασής τους. vielen Dank. Ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι είμαι λίγο έκπληκτος για τη γνωμοδότηση της Κομισιόν. Μας είπατε στην αρχή ότι έχετε πάρα πολλές αναφορές για το ίδιο θέμα, ότι λάβατε γραπτή θέση, ότι οι αναφερόμενοι ε, δεν έλαβαν κάποια απάντηση. Ε, μας φαίνεται εδώ ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και ότι θέλω να πιστήσω την προσοχή ότι κάθε πολίτη έχει δικαίωμα να απευθυνθεί σε αυτή την επιτροπή. Αν πείτε, αν λέτε εσεί ότι σε άλλε σε χώρες δεν έχετε τέτοια προβλήματα, δεν πρέπει αυτό να μα εμποδίζει να ασχοληθούμε με αυτέ εδώ τι αναφορέ. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με το ερώτημα του αν διαπράτεται παράβαση ευρωπαϊκού δικαίου, ε, παράβαση ε, νο, ε, για την, ε, της ελευθερίας εγκατάστασης, της οδηγίας παροχής υπηρεσιών του 2006 εσείς αντιθέτως μας λέτε για, τις, ε, για τα τέλη, για τις εισφορές των μελών, το οποίο είναι το πρόβλημα κατά την άποψή σας. Δεν βλέπω, ότι εγώ, ε, δεν βλέπω εγώ ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Άλλο είναι το πρόβλημα για το οποίο απευθύνονται εδώ οι αναφερόμενοι σε αυτήν εδώ την Επιτροπή και δεν ε, το λέω μόνο εγώ. Έχουν δικαίωμα οι άνθρωποι αυτοί να, κάνουν, να παρουσιάσουν την θέση τους. Και να σας πω επίσης ότι, η γραπτή ότι υπάρχει μια γραπτή νομοδότηση σε αυτήν την αναφορά την οποία έχουμε επεξεργαστεί και είναι καλό ότι το έχει κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι έχει ασχοληθεί δηλαδή με αυτήν την αναφορά τη δική μας, αλλά αρμοδιότητα των μελών αυτή τη Επιτροπής και αυτό που περιμένουν και, και οι αναφερόμενοι είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να να ασχολείται στα σοβαρά με αυτές τις αναφορές και να δει πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν σωστά και αντικειμενικά τα προβλήματα που εντοπίζονται. Εσείς λέτε τώρα ότι έχουν άδικο. Εγώ πιστεύω ότι έχουν δίκιο. Τουλάχιστον όμως εσείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μας δώσετε κάποια αιτιολογία, κάποια επιχειρήματα γιατί δεν έχουν δίκιο. Εδώ σε αυτή την αναφορά δεν έχετε λάβει καθόλου θέση η αναφορά που, στην οποία αναφέρεστε εσείς ε, γραπτά. Εσείς αναφέρεστε σε, σε διάφορες αναφορές στο παρελθόν, όχι όμως αυτήν εδώ, εδώ που συζητούμε τώρα. Οι άλλες οι ε, παρελθούσες αναφορές έχουν κάνει με άλλα πράγματα. Στη Γερμανία μπορεί το σύστημα μένει να είναι περίπλοκο των επιμελητηρίων, όμως υπάρχουν, αν κατάλαβα καλά, ε, τρία, διαφορετικά επιμελητήρια. Το επιμελητήριο των ελεύθερων επαγγελματιών, των γιατρών, των δικηγόρων κτλ. Υπάρχει το βιοτεχνικό επιμελητήριο και υπάρχει και το βιομηχανικό. Και γι' αυτό εδώ μιλάμε σήμερα. Όχι για το βιοτεχνικό. Δεν ανέφερε κανείς αυτό το πράγμα. Αναφερθήκαμε στους ελεύθερους επαγγελματίες. Και οι αναφορές που ε, για τις, στις, για οποίες ε, κάνατε λόγο έχουν να κάνουν άλλα πράγματα. Με το, εδώ έχουμε να κάνουμε με το βιομηχανικό και εμπορικό επιμελητήριο. Εμπορικό επιμελητήριο. Βιοτεχνικό και εμπορικό είναι διαφορετικά και νομικά διαφορετικά πράγματα. Και εμείς ως Επιτροπή έχουμε δικαίωμα και οι πολίτες έχουν δικαίωμα να πετήσουν από την Κομισιόν να ασχοληθεί ενεργά με το ζήτημα και να λάβει μια ε, θέση, να γνωμοδοτήσει για την ε, ελευθερία εγκατάστασης, για, την για τις παραβάσεις που έχουν συμβεί εδώ. Παραβάσεις και, για, ε, στην αρχή της δημοκρατίας, στο κάτω-κάτω. Δεν δεν αντιτίθεμαι στην ε, αυτοδιοίκηση των οργάνων αυτών, των επιμελητηρίων. Όμως, εάν υπάρχει ένα υποχρεωτικό σύστημα εγγραφής, εάν κάποιος υποχρεώνει, τότε πρέπει πραγματικά να δοθούν σαφείς, ξεκάθαροι νομικοί λόγοι και ξεκάθαρο πλαίσιο. Και όταν ένα επιμελητήριο με εμποδίζει να ασκήσω την επαγγελματική δραστηριότητα την οποία υποτίθεται προασπίζει και γι' αυτό πληρώνω, ε, έχουμε πρόβλημα. Εάν ε, ε, η οδηγία για την παροχή υπηρεσιών είναι λίγο σαφής, όπως για παράδειγμα στο παράδειγμα της Γερμανίας και της Αυστρίας, που, που επιτρέπεται να είμαι μέλος, που δεν επιτρέπεται να είμαι μέλος, πώς πρέπει να το επεξεργαστούμε αυτό με ορθό τρόπο. Και εδώ θέλω να πω σαφέστατα και ξεκάθαρα, να το πω για αγγλικά, back to sender. Το επιστρέφουμε σε εσά. Πάρτε πίσω αυτό που μας παρουσιάσατε, ξανασκεφτείτε το, δείτε την ε, αναφορά προσεκτικά, αυτήν εδώ, αναλύστε τι και μετά επανέλθετε. Και θα συμβούλευα να την εξετάσετε μαζί με την αναφορά από την Ελλάδα σχετικά με την ε, υποχρεωτική εγγραφή σε επιμελητήρια στην Ελλάδα. Ε, δεν μπορούσα δυστυχώς να την καταλάβω γιατί δεν μεταφράστηκε στα γερμανικά. Όμως πιστεύω ότι την επόμενη φορά μπορούμε να το βάλουμε στην ημερήσια διάταξη για να καταλάβουμε και την ελληνική περίπτωση, την ελληνική αναφορά και να δούμε να μπορούμε να ζητήσουμε μια σωστή επί της ουσίας και αντικειμενική αυτή τη φορά θέση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που να, ασχοληθεί με την περίπτωση της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας. Η... Ναι, η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα. Η Γερμανία και η Αυστρία είναι οι χώρες που έφεραν αυτήν την έκθεση. Στην Ισπανία είναι το αντίθετο αποφασίστηκε το αντίθετο και εγώ θα, ε, εμένα θα με ενδιαφέρε προσωπικά πολύ να μάθω για ποιου λόγους οι Ισπανοί κατήργησαν τις υποχρεωτικές εγγραφές και ποιε συνέπειε έχει αυτό. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το θέμα το αντιμετωπίζουμε, ναι, όντως, ως ε, η Γερμανία, την υποχρεωτική έγγραφη. Αυτό που δεν αναφέρθηκε μέχρι τώρα είναι ότι και τα βιομηχανικά επιμελητήρια έχουν αυτοδιοικητικά όργανα. Έχετε χιλιάδες μέλη τα οποία μπορούν να εξετάσουν αυτό το ζήτημα. Μπορούν να συζητήσουν όλα αυτά τα ζητήματα, τα προβλήματα που προκύπτουν από την υποχρεωτική εγγραφή στα επιμελητήρια. Μπορείτε να αναθέσετε και σε αυτούς στο κράτος. το κράτος μπορεί να απαιτήσει και αυτό κάποιες επιπλέον ενέργειες, ε, ε, κόστος, ε, αναθεώρηση, επανεξετάσεις. Υπάρχουν βιομηχανικά επιμελητήρια που πραγματικά είναι αξιοκατάκριτα. Υπάρχουν και άλλα όμω που δεν είναι. Υπάρχουν και άλλα που είναι αρκετά επιτυχή στο έργο του. Κάποια που πραγματικά αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των πολιτών. Κάποια που καθόλου. Είναι μια γερμανική ιδιαιτερότητα ε, αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες που προσφέρουν τα επιμελητήρια, που βοηθούν. Ε, αυτή τη συζήτηση την ξέρω πολύ καλά. Στη Γερμανία είναι θέμα που συζητιέται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το ερώτημα που προκύπτει από όλο αυτό είναι εάν υπάρχει αυτή η ελευθερία εγκατάστασης, εάν υπάρχει παράβαση στην ελευθερία εγκατάστασης και στην οδηγία για την ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Και αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Όμως ε, κλείνω, κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι να επαναλάβω ότι το βιομηχανικό επιμελητήριο είναι ένα αυτοδιοικούμενο όργανο και τα επιμελητήρια αυτά χωρίζονται σε διαφορετικούς τομείς ανάλογα με τα, επαγγέλματα. Έχουν πολύ διαφορετικές ε, αρμοδιότητες, ε, πολύ διαφορετικούς αριθμού μελών. Κάποιο έχει 60.000 μέλη, κάποιο έχει 3.000 μέλη για παράδειγμα. Ξέρω εγώ αυτά που έχουν λιγότερα μέλη. Για παράδειγμα στον ε, τομέα της εστίασης. Είναι πολύ διαφορετική. Τι είναι και η διαφορά στα μέλη, στον αριθμό των μελών που είπατε και πριν. Και το, όσο για το πόσο δημοκρατικά ενεργούν τα επιμελητήρια αυτά, πρέπει να ληφθούν πολλοί παράγοντες υπόψη. Οι ιδιαιτερότητες στη δομή. Φυσικά μπορούμε να τα αποκαλέσουμε μη δημοκρατικά και τον τρόπο λειτουργία το ΣΜΗ δημοκρατικό, όμω δεν φτάνει μόνο να κάνουμε γενικεύσεις. Πρέπει να δούμε τους επιμέρους τομεί και τις διαφορές και τις ιδιαίτερότητε και των τομέων αυτών και του γερμανικού συστήματο με τα επιμελητήρια. Να, αυτό που μας είπατε, 21 ψήφοι που είναι αναγκαίες για μία θέση κτλ. Κλείνω, κλείνω. Υπάρχουν αρμοδιότητες που έχει το κράτος, πράγματα που πρέπει να κάνει το κράτος, τα οποία αυτούς τους αυτοδιοικούμενους οργανισμούς, τα οποία θα αναφέρονται σε αυτούς τους αυτοδιοικούμενους ε, οργανισμούς, αυτά τα επιμελητήρια. Μπορούν να ασχοληθούν για παράδειγμα για το ζήτημα των υποχρεωτικών εισφορών, της κατάρτισης. Και αυτό που ακούσαμε σήμερα, αυτή η κριτική που ασκήθηκε για μένα, όπως ανέφερα, δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι κριτική όμως που πιστεύω ότι ασκείται σε συγκεκριμένα επιμελητήρια που έχουν κάνει συγκεκριμένα λάθη. Και το ζήτημα μπορεί να, γίνει και, μπορεί να είναι και πολιτικό. Εσείς λέτε ότι ενεργείτε για το, ε, προς το συμφέρον των ε, μελών σας. Και το ξέρω αυτό, το έχω ακούσει πολλές φορές. Υπάρχουν όμως τα μεγάλα ψάρια στη θάλασσα και τα μικρά ψάρια. Υπάρχουν άλλα συμφέροντα και υπάρχουν και συμφέροντα. Τα προβλήματα λοιπόν που εσείς μας φαίνεται εκτός μικροφώνου ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ. Θα παρακαλέσω τους επόμενους να μιλήσουν λίγο γρήγορα γιατί έχουμε να απασχοληθούμε και με μια ακόμη σημαντική ε, αναφορά. Επομένως παρακαλώ τον, ε, τους κυρίους στην Άρου και τον κύριο Χέφνερ να είναι λίγο σύντομοι. Ευχαριστώ. Θα συνοψίσω αυτά που είπε ο συνάδελφο Χέφνερ. Σύμφωνο μαζί του οι αναφερόμενοι θέλουν να καταργηθούν τα επιμελητήρια. Όχι, δεν θέλουν να καταργηθούν τα επιμελητήρια. Θέλουν να καταργηθεί η υποχρεωτική εγγραφή σε επιμελητήριο. Και πολλά από τα προβλήματα που συζητήθηκαν έχουν να κάνουν με το υποχρεωτικό τη εγγραφή. Εάν, εγώ, δεν είμαι υποχρεωμένο να συμμετέχω σε ένα επιμελητήριο, ε, δεν είμαι υποχρεωμένο, μπορώ να το κάνω εθελοντικά και να αποδεχτώ και εθελοντικά του όρου είναι διαφορετική όμως η κατάσταση όταν είναι κάτι υποχρεωτικό. Γι' αυτό λοιπόν Καταρχά θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που είπε ο συνάδελφος Χέφνερ. Η αναφορά αυτή να εξεταστεί στα σοβαρά και αντικειμενικά. Και η, και η αναφορά των ε, επιχειρήσεων αυτών. Εγώ θα έλεγα ότι αν ε, δεν ήταν επιχειρήσεις αλλά άνθρωποι θα έλεγα ότι υπάρχουν παραβιάσεις των, ε, της προσωπικής μου ελευθερίας. Αναφερόμαστε όμως τα επιχειρήσει. Στην, στον αγροτικό τομέα, για παράδειγμα, ισχύουν άλλα πράγματα. Αν είμαι ελεύθερος επαγγελματίας γεωργός, δεν είμαι υποχρεωμένος να συμμετέχω ε, σε επιμελητήριο, όμως αν έχω κάποια ε, ιδιαίτερη εταιρεία Γκέμπεχα για παράδειγμα, είναι, είναι το ζήτημα αρκετά περίπλοκο. Ανάλογα με ποια νομική μορφή έχει μια ε, εταιρεία πρέπει να έχει υποχρέωση ή όχι να συμμετέχει να εγγραφεί σε επιμελητήριο. Σαφώ, καθώ φαίνεται, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει διαφορετική νομοθεσία για τα επιμελητήρια. Κάποιε χώρε έχουν, κάποιε χώρε δεν έχουν, είδαμε. Δεν όμως πιστεύω ότι το πρόβλημα εδώ είναι οι αρμοδιότητες του επιμελητηρίου, αλλά το γεγονός ότι τα επιμελητήρια είναι οργανισμοί που έχουν μεν αρμοδιότητες, αλλά παρουσιάζουν και πάρα πολλά προβλήματα. Το πρόβλημα λοιπόν για μένα έγκυται στο υποχρεωτικό της εγγραφής σε επιμελητήριο. Εκτός μικροφώνου. Wenn Όπως ενημερώθηκα υπάρχουν και, οργανισμοί επιμελητηρίων σε ομοσπονδιακά επίπεδα, ενώσει ε, τοπικών επιμελητηρίων. Όμως γενικά συνοψίζοντας ε, μπορούμε να αφήσουμε, πιστεύω, συνιστώ μάλλον να αφήσουμε το θέμα ανοιχτό και να το αναλύσουμε παραπάνω και με τους νομικούς εμπειρογνώμονές μας να τους, να τους μεταφέρουμε αυτή την αναφορά. Δεν θα ήθελα εγώ προσωπικά να κλείσω αυτή την αναφορά αλλά να το εξετάσουμε και να το... γιατί πράγματι πιστεύω ότι δεν είναι και τόσο δημοκρατική η υποχρεωτική εγγραφή. Ε, ο κύριος Μποστινάρου. Μικρόφωνο, παρακαλώ, μικρόφωνο. Δεν έχει ανάψει το μικρόφωνο του ομιλητής. Είναι αληθές ότι οι κανόνες που διέπουν τα εμπορικά επιμελητήρια ανήκουν στην επικουρικότητα. Αυτό είναι αληθές. Αλλά εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Δεν πρόκειται για δημόσιες οντότητες που καλύπτουν κυβερνήσεις και ευθύνες κρατών. Πρόκειται για ιδιωτικές οντότητες ε, που ε, περιλαμβάνουν πρωταγωνιστές ιδιώτες δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε το κράτος για αυτά που κάνουν οι ιδιωτικές οντότητες. Ε, τρίτον, για μένα η απάντηση της Επιτροπής δεν είναι πλήρης, ε, δεν είναι περιεκτική, δεν είναι ολοκληρωμένη, διότι ένα θέμα δεν περιλαμβάνεται. Πρόκειται για αυτήν την υποχρεωτική υποχρέωση. Ε, μια, είναι περιορισμός της ελεύθερου ανταγωνισμού ή όχι. Είναι ένα θέμα που καλύπτει προβλήματα που σχετίζονται με προστατευτισμό ή όχι. Διότι όταν είναι κανείς υποχρεωμένος να πληρώσει ένα μεγάλο ποσό ως συνδρομή ε, για να γίνει μέλος ενός τέτοιου επιμελητηρίου, αυτό θα περιορίσει πάρα πολύ τις οικονομικές δυνατότητες και την ισότητα μεταξύ των αγορών. Και τέλος, ναι, να μείνει ανοιχτή η αναφορά θα καλούσα την Επιτροπή μας να στείλει το περιεχόμενο στην Ήτρε ε, διότι πρόκειται και για τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Θα πρέπει να εμπλέξουμε τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και ε, θα μπορεί ε, με βάση την αμοιβαιότητα η Γερμανία να αντιμετωπίσει το θέμα. Θα μπορούσαμε τότε να δούμε τι γίνεται όταν τόσες πολλές ισχυρές εταιρείες γερμανικές θα υποχρεωθούν να κάνουν το ίδιο στη χώρα μου, τη Ρουμανία ή σε άλλες χώρες. Νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα θέματα αυτά. Να ε, ε, μιλήσετε πάλι. Ε, Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ε, αυτό που ήθελα μόνο είναι πάρα πολύ σύντομα να μιλήσω για το τι πρέπει να κάνουμε και με τι πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Να το πω στο συνάδελφο. Αγαπητέ συνάδελφε Κοίτσμαν, Εσεί μα είπατε πολλέ φορέ ότι ξέρετε αυτή τη συζήτηση, Είδα σα είναι άγνωστη από τη Γερμανία, είναι πολιτικό το ζήτημα. Πρέπει να σα πω ότι ναι, το κόμμα σα ασχολείται με αυτό πραγματικά και είναι και διχασμένο για το ζήτημα αυτό. Ο συνάδελφό σα που ανήκει στην ίδια παράταξη έχει άλλη άποψη από εσά. Όλα αυτά είναι μια πολιτική συζήτηση εντό γερμανικών συνόρων που δεν πρέπει να μεταφερθεί εδώ. Εδώ μας έχει τεθεί ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα που αφορά ευρωπαϊκή νομοθεσία. Να το βλέπετε. Και εγώ θεωρώ αυτή την ε, σύνοψη σε δύο σελίδες της αναφοράς πάρα πολύ ε, ωφέλιμη. Τα βασικά ε, περιεχόμενα της αίτησης της αναφοράς αυτής είναι η παράβαση ευρωπαϊκού δικαίου και, της, και των δημοκρατικών μας αρχών. Όλα τα υπόλοιπα είναι, είναι πράγματα που αφορούν τη Γερμανία και είναι πολιτικές συζητήσεις και να τις κάνετε στο κοινοβούλιο σας Παρακαλούμε όμως εμεί εδώ πραγματικά επιγόντω την Κομισιόν να καταρτήσει μια νέα γνωμοδότηση για αυτά τα συγκεκριμένα σημεία. Όχι, μην, όχι τώρα για τους κτηνιάτρους, για τους ε, φαρμακοποιούς, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε πάντως προκύπτει, ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο, πρώτον η χρησιμότητα των επιμελητηρίων ανά την Ευρώπη, ε, δεύτερον ε, το κενό, ε, το νομικό που υπάρχει ανάμεσα στα διάφορα κράτη και αυτό ίσως θα πρέπει να απασχολήσει την ε, Επιτροπή οπωσδήποτε. Επομένως πρέπει να το δούμε με κάποιο τρόπο για να μην έχουμε τέτοιες μορφής ε, αντιφατικές στάσεις ανάμεσα στα κράτη με το καπέλο της επικουρικότητας. Προτείνω να την αφήσουμε ανοιχτή ε, παρόλο που κατανοώ την Επιτροπή στο ότι δεν μπορεί να δώσει απάντηση πέρα από το αν γίνεται παράβαση ή όχι του ευρωπαϊκού ε, τιμένου με την έννοια ότι δεν υπάρχει νομοθεσία που να ε, αντιβαίνεται αυτή τη στιγμή με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο. Επομένως, να αφήσουμε την πρόταση ανοιχτή, να, την, ε, να διαβιβάσουμε το ζήτημα στην Ήτρε και στην Γιούρη, προκειμένου να δουν αν μπορούν να καλύψουν αυτό το κενό. Επομένως, είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα το οποίο πιθανόν να το καλύψουμε στην πορεία. Ευχαριστώ. Ε, μια αναφορά από τον κύριο Ιβά Μαρτά ε, που είναι παρόν και θα μας παρουσιάσει ένα ζήτημα που έχει σχέση με ένα λατομείο στο οποίο η εταιρεία ζητάει άδεια να κατέβει σε αποθέματα ε, πορολίθου χαμηλότερα από την επιφάνεια του εδάφους. κύριε Μαρτέν, παρακαλώ να μας παρουσιάσετε την αναφορά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εισαγωγικά θα ήθελα να υπενθυμίσω αυτά τα όσα διευκρινίσατε. Όντως πρόκειται ε, για ένα λατομείο ασβεστόλιθου που έχει σκοπό να εμβαθύνει κατά 35 μέτρα επιπλέον πράγμα που θα έρθει να ε, συναντήσει δύο υπόγειους υδάτονες υδροφόρους ορίζοντες ε, και θα θέσει σε κίνδυνο αυτούς τους υδάτινους πόρους. Θα ρηπανθούν, η ποιότητά τους θα υποβαθμιστεί και θα μειωθεί και η ποσότητά τους. Προτού περάσω στα διάφορα σημεία τα οποία μας θέτουν προβλήματα, θα ήθελα να υπενθυμίσω ιστορικά την όλη διεξαγωγή. Καταθέσαμε το 2011 την αναφορά, παρουσιάστηκε μια πρώτη φορά τον Ιούνιο 2011 και ορισμένες ερωτήσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτές οι ερωτήσεις ε, υποβλήθηκαν στις γαλλικές αρχές. Δόθηκαν απαντήσεις, ένα σημείωμα από τις γαλλικές αρχές για, ως απάντηση στα διάφορα σημεία, σημεία τα οποία είχαν ως θέμα την μη συμμόρφωση προς τις ευρωπαϊκές αρχές. Λάβαμε την απάντηση στο τέλος του Μαρτίου και ε, από τις οργανώσεις μας εκπονήσαμε ένα έγγραφο απαντητικό αρκετά ε, ογκώδες ε, που διαβιβάσαμε στις αρχές του Ιουνίου στην Επιτροπή για να απαντήσουμε στο σημείωμα των αρχών σχετικά με τα διάφορα σημεία που είχαν αναφερθεί. Υπήρξε μια διαδικασία στην Γαλλία που έδωσε την άδεια αυτή η διαδικασία είναι μια διοικητική διαδικασία και η άδεια δόθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2010. Η σημερινή κατάσταση είναι ότι ο βιομήχανος Λαφάρ, Σιμέντα Λαφάρζ έχει την άδεια για να εμβαθύνει ε, το λατομείο ε, παρά τα διάφορα σημεία τα οποία έρχονται είναι παραβάσεις ε, των οδηγιών των κοινοτικών. Θα υπενθυμίσω τα σημεία που αναφέρομαι στο έγγραφο αυτό. Το έγγραφο αυτό αποτελείται από μια περίληψη συνοπτική τεσσάρων σελίδων που βασίζεται σε ένα παράρτημα που διευκρινίζει διεξοδικά τα διάφορα σημεία ε, και έχει και 29 αποδεικτικά έγγραφα που προέρχονται είτε από την έρευνα όταν αυτή έγινε είτε για τις περισσότερα, τα περισσότερα παιδοκτικά στοιχεία από πρόσθετα στοιχεία τα οποία εκπονήσαμε και ανακαλύψαμε διάρκεια των μελετών. Υπάρχουν δύο μεγάλα σημεία τα οποία αμφισβητούμε. Πρώτον είναι η υποβάθμιση των υπογείων υδάτων και των επιφανειακών υδάτων, διότι να βγουν στον αέρα αυτές τα φρεατικά ύδατα απειλούνται από ρήπανση. Έχω ένα παράδειγμα, παρόλες τις δηλώσεις καλής θέλησης, παρατήρησα ότι για ορισμένες αναφορές έχει λεχθεί ότι δεν αρκούν οι καλές προθέσεις. Το 2007, παρόλη την καλή θέληση του βιομήχανου, υπήρξε μια ρήπανση με πυρίτιδα σιδήρου στον ποταμό που βρίσκεται κοντά στο λατομείο και είχαμε μια μεγάλη θνησιμότητα ψαριών. Ακολούθησε μια έρευνα. Συνεπώς έχουμε ένα παράδειγμα συγκεκριμένο κινδύνου ρήπανσης που γίνεται πραγματική ρήπανση. Αυτό το αποδεικτικό έγγραφο προσαρτήθηκε στο ε, φάκελο που διαβιβάσαμε στην Επιτροπή Αναφερών και αναφέρουμε λοιπόν αυτό τον κίνδυνο ρήπανση και την παράβαση σε σχέση με τις εγγυήσεις που πρέπει να δίνονται σε συμμόρφωση προς τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι ρήπανση με τα χημικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στο λατομείο, στο σημείωμα των γαλλικών αρχών που μας διαβιβάστηκε το Μάρτιο, αναφέρεται ότι δεν υπάρχει κανένα ε, χημικό που χρησιμοποιείται στο λατομείο. Αυτό είναι αναλυθές, διότι για να γίνει η εμβάθυνση χρησιμοποιούν εκρηκτικά και τα εκρηκτικά αυτά τοποθετούνται εντός του βράχου για να χρησιμοποιηθούν. Υπάρχει λοιπόν, έρχονται σε ε, οι φρεατικές, ε, τα φρεατικά ύδατα έρχονται σε επαφή λοιπόν με, τα, με τις χημικές ουσίες στο έγγραφο των αρχών των γαλλικών υπάρχει ένα όριο που ορίστηκε για τις απορρίψεις ατράκων που ορίστηκαν με 85 λίτρα απόρριψη κατά ημέρα, είναι ένα ανώτατο όριο βλέπουμε εδώ τις καλές προθέσεις του βιομηχάνου, αλλά πώς μπορεί να δοθεί μια άδεια με μια άδεια απόρριψης ε, στην φύση 85 λίτρων την ημέρα υδρογονανθράκων. Αυτό είναι ε, πάρα πολύ σημαντικό και όταν δούμε τους στόχους, ε, τους ποιοτικού ε, για το είδωρ με στην οδηγία, την πλαίσιο για το είδωρ, αυτό έρχεται σε αντίφαση και είναι μία παράβαση και είναι απαράδεκτο. Όλες οι μελέτες που έγιναν για να δοθεί αυτή η άδεια έγιναν στο, ακριβώς στο στην περίμετρο του λατομείου. Αλλά έχουμε λάβει από τότε ορισμένες πληροφορίες που έδειξαν ότι υπάρχουν επιπτώσεις πέραν της περιμέτρου, δηλαδή στις δύο ζώνες Natura 2000 που είναι όμορες του λατομείου, που βρίσκονται σε λιγότερη απόσταση από 300 μέτρα. Υπάρχει ένας υγροβιότοπος που θα επηρεαστεί από την αποξήρανση των υδάτων και θα έχουμε κατά συνέπεια εξαφάνιση της χλωρίδας και επανίδας που ε, σχετίζεται με τον υγροβιότοπο. Είναι απαράδεκτο σε μια μελέτη να εστιαζόμαστε μόνο στην δικητική περίμετρο του ορυχείου και να μην εξετάζουμε το ε, περιβάλλον γύρω από το, από το λατομείο, δηλαδή στα 50 μέτρα. Δεν ξέρω ότι δεν είναι τόσο μακριά αυτή, αυτός ο υδροβιότοπος. Επίσης, οι οργανώσεις μας θέλησαν στο έγγραφο που διαβιβάσαμε να διευκρινίσουν ορισμένα άλλα σημεία πλαισίου. Θέλουμε να θέσουμε στη διάθεση της Επιτροπής ορισμένες πληροφορίες σχετικά με συνδέσεις που υπάρχουν, στενές σχέσεις ανάμεσα στον βιομήχανο και διάφορες οργανώσεις. Οι οργανώσεις αυτές οι οποίες κάνουν τώρα τις αξιολογήσεις αντικτύπου και είναι απαράδεκτο να ανακαλύπτουμε ότι οι επιδοτήσεις από τον βιομήχανο δόθηκαν σε οργανώσεις που επιφορτίστηκαν από το κράτος να τοποθετήσουν μετρητές ε, του αντικτύπου ε, ε, του, περιβαλλοντικού. Έχουμε λοιπόν αποδεικτικά στοιχεία στο, στο φάκελο και θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε το σύνολο αυτών των πληροφοριών. Εν κατακλείδη, βλέποντας όλα αυτά τα σημεία, θεωρούμε ότι υπάρχει παράβαση των οδηγιών πλαισίων για το είδωρ και για τον λόγο αυτό διαβιβάσαμε το έγγραφο που είναι μια απάντηση στο σημείωμα των γαλλικών αρχών ούτω ώστε να σας γνωστοποιήσουμε ορισμένες λεπτομέρειες που δεν θα αναφέρω εδώ ε, ενδελεχώς αλλά που μπορείτε να βρείτε ε, στο έγγραφο που βρίσκεται στο φακελό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. σας ευχαριστώ από την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εκπροσωπώ την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Επιτροπής και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι όπως αναφέρθηκε είχαμε την αναφορά αυτή ήδη το 2010, την κοινοποιήσαμε στην Επιτροπή σας εκείνη την εποχή, οι πληροφορίες εκείνη την εποχή που μας δόθηκαν δεν ήταν ε, ε, μια βάση σχετικά με τις οδηγίες το 2010. Υπήρξαν δημόσιες διαβουλεύσεις εκείνη την εποχή ε, και οι γαλλικές αρχές ε, οδηγήθηκαν σε μια απόφαση από τότε και πρόσφατα λάβαμε νέες πληροφορίες σχετικά με την αναφορά αυτή. Τώρα, όπως ακούσαμε, οι γαλλικές αρχές επίσης έδωσαν άδεια για την εμβάθυνση του λατομείου και από ό,τι καταλάβαμε από τον αναφέροντα σε αυτήν την περίληψη που ανέφερε, την περίληψη της, ε, των προσθέτων πληροφοριών, οι αναφέροντες έχουν ε, διάφορα προβλήματα ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ε, προβλήματα ρήπανσης υδάτων, επιφανειακών υδάτων, ε, υπογείων υδάτων. Επίσης υπάρχουν και οι ζώνες Natura 2000. Ε, Υπάρχει η νομοθεσία περί διατήρησης της φύσης που και επίσης ε, οδηγία περί αξιολόγησης περιβαλλοντικής στρατηγικής ε, που ε, νομίζω ενδιαφέρονται από την, τις νέες πληροφορίες που λάβαμε. Όλες οι πληροφορίες δεν μας έφτασαν, ήρθαν μερικές πολύ πρόσφατα λόγω των διαφόρων περιβαλλοντικών ε, τομέων χρειάζεται συντονισμός ε, με τους συναδέλφους ε, Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και είναι πρόωρο να εξαγάγω συμπεράσματα σχετικά με το πραγματικό πλαίσιο αυτό το οποίο μπορώ να πω τώρα είναι ότι όταν θα λάβουμε όλα τα έγγραφα αυτά, τα 29 έγγραφα που αναφέρονται εδώ, η Επιτροπή θα εξετάσει εντελεχώς όλες αυτές τις πληροφορίες και και η Επιτροπή θα εξετάσει αν όλοι η νομοθεσία ικανοποιείται και αν δεν υπάρχει παράβαση με βάση αυτές τις νέες πληροφορίες και αν κριθεί αυτό απαραίτητο θα ζητήσουμε στους γαλλικές αρχές πρόσθετες διευκρινήσεις, θα τους θέσουμε νέες ερωτήσεις για νέες πληροφορίες για να μπορέσουμε να καταλήξουμε για το θέμα αυτό. Και θα, θα ενημερώσουμε σχετικά την Επιτροπή αυτή. she's speaking. ich, sage meine, ich, äh, also ich sagen. Μάλιστα. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι η Κομισιόν δεν μπόρεσε να εξετάσει όλες τις πληροφορίες, γι' αυτό η αίτηση πρέπει να παραμείνει ανοιχτή. Παρακαλώ όμως ε, να ενημερώνεται, να ζητάει η Γραμματεία από την Κομισιόν ε, τακτικά για τακτικές ενημερώσεις σχετικά με την πορεία αυτής της αναφοράς, έτσι ώστε να μην ξεχαστεί. Ο αναφερόμενος εδώ έχει έχει ε, καταβάλει τις αιτήσει του, τις ερωτήσεις του για... και αξίζει μια απάντηση. Γι' αυτό και συνιστώ να την κρατήσουμε ανοιχτή για να συμπληρωθούν και οι πληροφορίε που λείπουν από την Κομισιόν. Μάλιστα, προφανέ είναι ότι πρέπει να μείνει ανοιχτό το ζήτημα και πραγματικά εξεπλάγει όταν έμαθα ότι η Κομισιόν είχε λάβει τις πληροφορίες εδώ και πολύ καιρό. και μπορούσατε να τις ε, μεταβιβάσετε σε κάποιον. Όμως τώρα εσείς μας λέτε ότι το λάβατε μόλις την Παρασκευή και αυτό μας προκαλεί κάπως έκπληξη. Τέλος πάντων όμως. Μπορούμε να το δούμε αυτό ίσως τον Οκτώβριο ανάμεσα σε δύο συνεδριάσεις αν μπορούμε να πάμε εκεί και να το δούμε με τα μάτια μας, γιατί είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Εάν αληθεύει, φυσικά και είναι μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Και εγώ πιστεύω ότι το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό. Ε, Α, κύριε Βοστινάρου, συγγνώμη, παρακαλώ. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Είναι κάτι σαν τεζαβή. Δηλαδή, πώς να εμπιστευτούμε στην ε, περιβαλλοντική μελέτη αντικτύπου όταν γίνεται από τους φίλους των φίλων μου. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα αυτό που συνεχώς ε, επανεμφανίζεται και δεν έχει επιληθεί ακόμη. Δεύτερο. Δεν λέγεται ούτε μία λέξη για την αναγκαιότητα αξιολόγησης των σωρευτικών αποτελεσμάτων, ε, γιατί έχουμε και την οδηγία για τα ύδατα, αλλά έχουμε και τη ρήπανση των ε, υπόγειων υδάτων αλλά και των επιφανειακών υδάτων και όπως είπατε χρειάζεται μια στρατηγική μελέτη αντικτύπου περιβαλλοντική. Εδώ έχουμε μόνο την περιβαλλοντική μελέτη αντικτύπου όπως είπε ο αναφέρον που προετοιμάστηκε από τους φίλους των φίλων μου. Και τέλος, να προτείνω να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και κατόπιν να εξετάσουμε τη δυνατότητα να μεταβούμε επιτόπου, να δούμε την πραγματικότητα και να ζητήσουμε φυσικά νέα αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί από το 2010 είχαμε χάσει μόνο, έχουμε χάσει μόνο δύο χρόνια. Βεβαίω θα κρατήσουμε την ε, υπόθεση, την αναφορά ανοιχτή. Ε, η Επιτροπή θα πρέπει να μας απαντήσει, παρακαλώ, να μας απαντήσει σχετικά με ένα έγγραφο που έχουμε στείλει για την υπόθεση το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε πριν από το τέλος Ιουλίου προκειμένου να δούμε πώς θα κινηθούμε στη συνέχεια αν πρέπει να κάνουμε μια ε, fact finding mission ή όχι αλλά σε κάθε περίπτωση το ζήτημα είναι απολύτως επίγον και πρέπει να ξεκαθαριστεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θα θέλατε να πείτε κάτι, κύριε, ο θα θέλατε να πείτε κάτι. Είναι προφανέ ότι αν χρειάζεστε συμπληρωματικέ πληροφορίε, είμαστε στη διάθεσή σα για να τι διαβιβάσουμε είτε τα έγγραφα που έχουν ήδη σταλεί ή άλλε πρόσθετε πληροφορίε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και αν θέλετε να έρθετε επί τόπου... Τι Είπατε κάτι? Okay. I'll speak English now. Uh, to, to keep... Λοιπόν, αιτήματα να διατηρήσουμε ανοιχτές τις αναφορές για το τμήμα Β. 22 της κυρίας 24 κύριο 33 κυρία Βαλεάν, 35 κυρία Άουκεν, 63 κυρία Άουκεν, 74 κυρία Ματσόνη και 79 και πάλι η κυρία Άουκεν. Ωραία, σας ευχαριστώ όλους για την υπομονή σας και σας ευχαριστώ που παρευρεθήκατε εδώ.